Bueno, buenas tardes. Καλησπέρα σας. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε λίγο καθυστερήσει. Καταρχήν, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους που θα συμμετέχουν ως εισηγητές σε αυτή τη δημόσια κρόση και επίσης ε, τους παρευρισκόμενους και θα σας εξηγήσω πολύ σύντομα πώς ε, θα υλοποιήσουμε αυτή την ακρόση. Καταρχήν και όπως ε, πάντα θα προσπαθήσουμε να σεβαστούμε τους χρόνους γιατί κάποιος τελικά δεν θα καταφέρει να πάρει το λόγο. Καταρχήν θα πάρει το λόγο η κυρία ρόντου, που είναι η εισηγήτρια για το βασικό κανονισμό για τη μεταρρύθμιση της ε, κοινωνικής Πολιτική και κατόπιν ο κύριο Ερνέστο Πένας, ο οποίο είναι διευθυντή τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΜΑΡΕ για μια εισαγωγή, πέντε λεπτά ο καθένα. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το πρώτο πάνελ. Έχουμε δύο πάνελ, ε, όπως γνωρίζετε στην ακρόαση αυτή. Το πρώτο ε, οι πρωταγωνιστές μιας περιφερειοποιημένης κάλπ και το δεύτερο σχετικά με τους στόχους ε, και τα μέσα για μια περιφερειοποιημένη κοινή πολιτική. Στο πρώτο πάνελ θα έχουμε πέντε ομιλητές, τέσσερις παρεμβάσεις, δέκα λεπτών και η τελευταία παρουσίαση από τον κύριο Μπαριόλα εξ όλων των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, περίπου 30 λεπτά θα μιλήσει και κατόπιν θα υπάρχει μία συζήτηση προκειμένου και οι υπόλοιποι βουλευτέ να μπορούν ε, να συμμετέχουν και να θέσουν τι ερωτήσει που θεωρούν σκόπιμε σε κάθε έναν από του προσκεκλημένου. Μία ώρα προβλέπουμε γι' αυτό. Και περίπου στις 5 και 4 και 20 θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο πάνελ. Ε, θα ακολουθήσουμε την ίδια δομή. Εδώ έχουμε δύο παρεμβάσεις, 10 λεπτών καθεμία. Και κατόπιν θα ξεκινήσει η συζήτηση για 40 λεπτά περίπου με τελική παρέμβαση με συγχωρείτε της κυρίας Ρόντουστ για να ολοκληρώσουμε και στην προκαθορισμένη ώρα. Αν κάποιος τώρα δεν θέλει να σχολιάσει, νομίζω ότι θα δώσουμε το λόγο καταρχήν στην κυρία Ρόντουστ για 5 λεπτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ως εισηγήτρια για την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής θα ήθελα πρώτα να σας καλωσορίσω όλους και όλους. Χαίρομαι που έχουμε κοντά μας τόσους εμπειρογνώμονες από τους διαφόρους τομείς που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Εμείς στην Επιτροπή Αλληλεία συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε την περιφερειοποίηση. Βέβαια, οι απόψεις μας διήστανται σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες και μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε. Ωστόσο, όλοι θέλουμε να λαμβάνονται περισσότερες αποφάσεις επιτόπου με περισσότερη συμμετοχή των αλλιών. Δηλαδή, μια πολιτική η οποία να, την οποία να συνδιαμορφώνουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και όχι μια πολιτική που να υπαγορεύεται άνωθεν από τις Βρυξέλλες. Υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ε, εξηγηθεί και με ένα μη έγγραφο. Στο ίδιο το νομικό κείμενο διαλαμβάνονται οι ρόλοι των διαφόρων φορέων στα διάφορα επίπεδα. Και αυτό θέλουμε εμεί να το βελτιώσουμε. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερε αρμοδιότητε να δοθούν στο περιφερειακό επίπεδο, υπό δύο όμω όρου. Πρώτα, πρέπει να είναι διασφαλισμένο ότι οι στόχοι τη κοινή ελευθερική πολιτική θα επιτευχθούν. Δεύτερο, η περιφερειοποίηση θα πρέπει να είναι νόμιμη, δηλαδή συμβατή με τι ευρωπαϊκέ συνθήκε. Ω Επιτροπή Αλία έχουμε φτιάξει ένα κατάλογο ερωτήσεων των οποίων έχουμε υποβάλει. Με τι ερωτήσεις αυτές επιθυμούμε να βολιδοσκοπήσουμε εάν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στην περιφερειοποίηση από ό,τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δε νομικοί μα εμπειρογνώμονε επεξεργάζονται τώρα τι απαντήσει του. Εκτό αυτού, στο έγγραφο εργασία έχω κάνει ορισμένε προτάσει όπω μια δεσμευτική γνωμοδότηση των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, βέβαια με πιο δίκαιη σύνθεση τα συμβούλια αυτά. Οι χώρε μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την υποχρέωση όταν θα ψηφίζουν και εκδίδουν τα περιφερειακά μέτρα να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ζητώ επίσης βελτιωμένο ελεγκτικό μηχανισμό ώστε να εφαρμόζεται καλύτερα η κοινή στόχη και να μην ανησυχούμε εδώ εμείς στις Βρυξέλλες. Αναμένω με μεγάλη ανυπομονησία και ενδιαφέρον την ακρόαση και αναμένω βεβαίως τις σημαντικές προτάσεις και συστάσεις που θα υποβάλλετε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρόντους. Θα ακούσουμε τώρα τον Ενέστο Μπένιας από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Και εμείς ε, συμφωνούμε απόλυτα σε σχέση με τα αίτια, τα κίνητρα της πρότασής μας για την περιφερειοποίηση. Πρόκειται για να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη μικροδιαχείριση των Βρυξελών, δηλαδή το χαρακτήρα από πάνω προς τα κάτω που δείχνουν πολλές από τις πολιτικές για την αλία και έτσι λοιπόν η περιφερειοποίηση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσπάθεια επανεθνικοποίησης της κοινής πολιτικής αλλά για να βρεθεί ένας τρόπος για να να λαμβάνονται τα, ε, οι αποφάσεις για τα πιο τεχνικά μέτρα ε, από όσους ε, είναι πρωταγωνιστές σε τοπικό επίπεδο. Προτείνουμε ένα σύστημα η Επιτροπή δεν προσπαθεί να δώσει όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργούσαν ε, όλα τα σταδίες διαδικασίας και έχουμε δύο πολύ καλούς λόγους γι' αυτούς. Αναφερθήκαμε ήδη στον ένα πάρα πολλές φορές και πρόκειται για τη δυσκολία, για τη νομική βάση της Λίκης ε, Μπορούμε να πάμε πιο μακριά για να ε, τυποποιήσουμε, να επισημοποιήσουμε μηχανισμούς περιφερειακής συνεργασίας. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος και για μας είναι πολύ σαφές ότι η περιφερειοποίηση πρέπει να είναι μια σταδιακή διαδικασία όπου δεν προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα παντού από την πρώτη μέρα, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία εκμάθησης, ε, όπου ξεκινάμε από συγκεκριμένε περιπτώσεις και από εκεί και πέρα θα αναπτύξουμε μεθοδολογίες, πρακτικές για το πώς θα λαμβάνουμε αποφάσεις σε περιφερειακό επίπεδο και πάντοτε θα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό όποια και είναι η νομική βάση, από την ε, καλή βούληση των κρατών μελών να συνεργαστούν στα πλαίσια μιας περιοχής ή ενός ε, είδους αλίας. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα εκούσιο σύστημα που από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει βούληση από τα κράτη-μέλη, τα ενδιαφερόμενα μπορούν να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη λήψη αποφάσεων περιφερειακού χαρακτήρα. Και από εκεί και πέρα η ιδέα να θεσπίσουμε πολύ συγκεκριμένες ε, κνήσεις, ε, προδιαγραφές για το πώς θα γίνει αυτό όχι μόνο είναι δύσκολο νομοθετικά, είναι και αντιπαραγωγικό. Γιατί μία αποκεντρωπημένη εστίαση της πολιτικής με ένα μεγάλο βάρος των κρατών μελών και των πρωταγωνιστών επιτόπου, θα, εφόσον θέλουμε αυτό, θα ήταν ε, ε, αντιπαραγωγικό να το καθορίσουμε σε κάθε λεπτομεριά του από τις Βρυξέλλες. Δεν θέλουμε να έχουμε μικροδιαχείριση από τις Βρυξέλλες για το πώς θα λάβει η χώρα αυτή η περιφοριοποίηση και πριν από τα τέλη του έτους θα υπάρχει πρόταση της Κομισιόν, παραδείγματος χάρη, ε, και αποτελεί παράδειγμα αυτό, Πρόεδρε, για να καθορίσουμε ε, την εξάλληψη των απορριψεών στο Σκάγκερα και και αυτό γιατί υπάρχει ε, υποστήριξη από τις τρεις χώρες, από την Δανία και τη Σουηδία, μαζί με τη Σουηδία, για να λυθούν συγκεκριμένα μέτρα και κατόπιν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε στην νομοθεσία τη Ένωση να απαγιώσουμε ότι δύο κράτη-μέλη με μία τρίτη χώρα μέσω μία συνεργασία χωρί κανόνε, δηλαδή στην πράξη το κάνουν, δεν χρειάζονται την Κομισιόν να του πει πώ θα το κάνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα για το πώ μπορούμε να προωθήσουμε την περιφερειοποίηση. Από εκεί και πέρα, αυτό που χρειάζεται να βάλουμε στο βασικό κανονισμό της μελλοντική κάλπα ε, δεν είναι λεπτόμερείς οδηγίες για το πώς θα υλοποιηθεί, αλλά μια ευρεία νομική βάση που να επιτρέπει όταν ξεκινούν ε, οι εμπειρίες στα πράγματα της περιφερειοποίησης, τα κράτη-μέλη να μην αντιμετωπίζουν ε, νομικά εμπόδια, δηλαδή να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν το προβλέπει ο βασικός κανονισμός ή το εμποδίζει. Περί αυτού πρόκειται, Πρόεδρε. Πιστεύω λοιπόν ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε μία μικροδιαχείριση για να έχουμε ακριβώ μία πλήρω αποκεντρωμένη εστίαση. Και στα πέντε λεπτά θα ήθελα να απαντήσω και στι δύο ερωτήσει που τίθενται από την κυρία Ρόντουστ. Καταρχήν, ο ρόλο των Περιφερειακών Οργανωτικών Συμβουλίων. Να επιβεβαιώσω ότι για την Κομισιάν είναι πάρα πολύ σημαντικό η εστίαση των ε, αποκεντρωμένων αποφάσεων ε, να γίνεται με μηχανισμούς διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι τα ΡΑΚ και τα Περιφερειακά Γνωματικά Συμβούλια πρέπει να δραματίσουν ένα ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων και σε σχέση με τους μηχανισμούς ελέγχου. Να επενθυμίσω ότι όλες οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Κομισιόν στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου της ε, Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλίας ε, προ την κατεύθυνση της περιφερειοποίησης του ελέγχου. Τώρα, τα προγράμματα ελέγχου τα οποία συντονίζει η υπηρεσία στο Βίγκο ήδη έχουν προσαρμοστεί στην περιφερειοποίηση και ε, θέτουν εστίαση στην νομική βάση που θα θετηθεί και σε κάποιους μηχανισμούς περιφερειακού περιφερειακούς μηχανισμούς ελέγχου. Έτσι λοιπόν κυρία Ρόντου, το θέμα της περιφερειοποίησης χάρη στην δραστηριότητα της υπηρεσίας ελέγχου ήδη ε, υπάρχει και έχουμε πλήρη περιφερειοποίηση. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. On the legal basis question... Ευχαριστώ για το θέμα της ε, νομικής ε, βάσης. Ε, μας είπε η νομική μας υπηρεσία, το άρθρο 2 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ρήτα ότι δίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσει σε ένα κράτος μελός να επιτελέσει εξ ονόματός της σε κάποιες δραστηριότητες, υποθέτω και ίσως αυτό προκύψει με μεγαλύτερη σαφήνεια κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Υποθέσαμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει το πλαίσιο της κοινή και ορισμένε δράσει, στα πλαίσια αυτή θα ανατεθούν ε, σε επίπεδο καθημερινής διαχείρισης στα κράτη-μέλη. Εγώ είχα καταλάβει ότι υπήρχε νομική βάση. Ε, σίγουρα θα διευκρινιστεί το θέμα εν ευθέτω χρόνο. Θα περάσουμε τώρα στους ε, ομιλητές για το πρώτο πάνελ. Ε, είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί ε, τη περιφερειοποιημένη κοινή αλληλευτική πολιτική. Θα δούμε τον ορισμό, το ρόλο, τα καθήκοντα ε, καθενό, τα οικονομικά μέσα που υπάρχουν. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Γκρέγκορ Ζόμποργκ που ανήκει στην Ένωση Ελλήνων της Πολωνίας. Ε, καλωσορίσατε και σας δίνω το λόγο. Thank Szanowni Państwo, jestem rybakiem od 30 lat. Posiadam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ασχολούμαι με την αλληλεία εδώ και 30 χρόνια. Έχω ένα σκάφο σε μήκου 17 ε, μέτρων. Ε, το κλονόμισα από τον πατέρα μου που ήταν επίσης ψαράς και θα ήθελα και εγώ να μεταβιβάσω στο γιο μου με τη σειρά μου και το σκάφο και την εμπειρία μου για να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση. Όλα αυτά βεβαίω εξαρτώνται από τι αποφάσει που θα λάβετε εσεί. Ελπίζω να είναι δυνατόν η περιφερειοποίηση. Πρέπει να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία τη μεταβίβαση μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτικής πολιτική. Προ το παρόν όμω, ε, είναι μυστηριώδη, ενηγματική αυτή η περιφερειοποίηση. Δηλαδή δηλώνεται από όλου ότι επιθυμούν να την εφαρμόσουν, αλλά όταν ασχολούμαστε με την πρακτική εφαρμογή διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πρακτικά κολλήματα, συγκεκριμένα περίπλοκοι κανόνε που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης περίπλοκη κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να διαχειριστούμε ορθά του πόρου, χρειαζόμαστε ευελιξία και δυνατότητα ταχεία λήψη αποφάσεων, Όμω το γραφειοκρατικό σύστημα όπω έχει σήμερα δεν το επιτρέπει αυτό. Ε, πολλά πλεονεκτήματα θα απορρέουν από μια ταχεία εφαρμογή της περιφερειοποίησης ως προς ε, την ε, χρήση όλων των αλληλευτικών αποθεμάτων στις διάφορες θελάσσιες λεκάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αναμφίβολο και υπάρχει συμφωνία από αυτού. Οι αλληλείς, οι αρμόδιοι οργανισμοί, οι επιστήμονες συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε αυτή την περιφερειοποίηση. Σήμερα όμως ζούμε ένα πραγματικό φιάσκο της κοινή κοινή αλληλευτικής πολιτικής με τη μορφή που έχει μέχρι στιγμής. Ε, Μία έκφανση ε, αυτής της αποτυχίας είναι οι ανεύθυνες δράσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την προσπάθεια μεταρρύθμισης κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Λοιπόν, η περιφερειοποίηση λόγω αυτής της αποτυχίας είναι σημαντικότατο εργαλείο για να ορθοποδήσει η ευρωπαϊκή αλία και για να ε, καταπολεμήσουμε τις παθογένειες που υπάρχουν σήμερα στον κλάδο, ούτως ώστε οι αλίες και εγχώριες κοινότητες ε, να καταφέρουν να ξεφύγουν ε, και να βρουν μια εναλλακτική λύση ως προς τις πλημελείς προτάσεις που έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Ε, πλέον κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη εφαρμογής αρχής περιφερειοποίησης στην αλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που συζητείτε είναι ο χρόνος, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής καθώς και η έκταση ε, της περιφερειοποίησης. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρία γίνεται όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη γίνεται η περιφερειοποίηση. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει διαρμοδιότητε στον τομέα αυτό, αλλά όσο λιγότερε έχει, τόσο καλύτερο, τόσο, σε τόσο καλύτερη κατάσταση θα βρίσκονται και τα αχθή αποθέματα και οι ε, επαγγελματίε του κλάδου. Ε, σήμερα ε, κανείς δεν είναι δηλωμένος εχθρός ε, της περιφερειοποίησης της αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι μάλλον οι λεπτομέρειες, εφαρμοστικές λεπτομέρειες της νέας αυτής κατεύθυνσης. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να επικεντρωθώ στις παρατυπίες, στις παθογένειες που παρατηρούνται στο κλάδο αυτό και πιο συγκεκριμένα στην Βαλτική θάλασσα η παθογένεια αυτή είναι απότοκος του ότι λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, μέχρι ε, τούδε ε, στην, ε, στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και δεν υπάρχει επαρκής σύμβολη των αρμόδιων εθνικών οργανισμών, των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων και των επαγγελματιών του κλάδου. Ελπίζω ότι με τη σημερινή ακρόαση για την περιφερειοποίηση θα βελτιωθεί η κατάσταση όχι μόνο στη Βαλτική αλλά σε όλες τις λεκάνες ε, της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής την αλία στη Βαλτική θάλασσα ισοδυναμεί με παράταση της του προγράμματος της Διεθνούς Επιτροπής Αλίας για τη Βαλτική Θάλασσα. Αυτή η Επιτροπή ρύθμιζε την αλία στη Βαλτική πριν από το 2004. Από το 2004 και μετά η Βαλτική έγινε εσωτερική θαλάσσια λεκάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξελίξεις δυστυχώς δεν είναι θετικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς ε, ακολούθησε άκρητα και αβασάνιστα την γραμμή αυτή ε, της Διεθνούς ε, Επιτροπής για τη διαχείριση της αλίας. Στη Βαλτική έχουν γίνει διάφορες απόπειρες από πλευράς Πολωνίας να επηρεάσουμε την κατάσταση, αλλά μάταια στην ε, Βαλτική απουσιάζουν ε, σχεδόν παντελώς ε, οι έλεγχοι της Αλίας για ορισμένα μόνο κράτη, αλλά αντίθετα δέχονται τα πειρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαρκώς. Για τους ελέγχους και τα κράτη που υφίστανται αυτούς τους ελέγχους υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στους αρμόδιους ελεγκτικούς οργανισμούς. Μπορείτε λοιπόν να διαπιστώσετε ότι σε κάποια κράτη δεν γίνονται ποτέ έλεγχοι και συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή ε, πριν την 1η του 2004. Μεταξύ των ε, τότε και τώρα πρακτικών νομίζω θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος στα εξή. πρωτον Πρώτον, Κάποια κράτη-μέλη θέσπισαν ε, εθνικούς εγχώριους κανόνες που επιτρέπουν σημαντική υπέρβαση των ποσοστώσεων του βακαλάου. Το αιτιολογείται από τις ιδιαίτερα χαμηλές ποσοστώσεις ε, που χορηγήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποια κράτη. Ε, σημειώνεται λοιπόν σημαντική υπέρβαση των ποσοστώσεων ε, και οι εκθέσεις που κατατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Διεθνή Επιτροπή για Διαχείριση ελεία στη Βαλτική είναι μαγειρεμένες. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Ε, δεν μπορούμε ως εκ τούτου να αξιολογήσουμε σε ποια επίπεδα βρίσκονται τα αποθέματα και άρα δεν έχουμε τη σωστή βάση για να αποφασίσουμε για την κατανομή των ποσοστώσεων για τα επόμενα έτη. Τον Ιούλιο του 2011 καταθέσαμε μια επίσημη καταγγελία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε δεν αντέδρασε καθόλου. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα, η κατανομή των ποσοστώσεων για το Σολομό ανάσκαφος. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη προκύπτει από τα στοιχεία ότι δεν περιορίστηκε η αλία του Σολομού και όπως και για τον Μπακαλιάρο ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε τα αποθέματα και να χορηγηθούν οι ποσοστώσεις επί τη βάση αυτών των στοιχείων. Ε, τρίτο πρόβλημα, η υπεραλίευση των πελαγικών ειδών. Κανένας ούτε ποιοτικός ούτε ποσοτικός έλεγχος δεν επιτελείται και έτσι καταστρέφεται ολόκληρη η τροφική αλυσίδα την ε, Βαλτική. Η... Ατελείς αυτή η διαχείριση στη Βαλτική σχετίζεται επίσης ε, με τους κανόνες που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα ε, η βάση μιας πολιτικής απόφασης ε, καταρτίστηκε ένα πολυετές ε, σχέδιο για την αποκατάσταση του αποθέματος του Μπακαλιάρου στην Βαλτική. Θεσπίστηκε ακριβώς την στιγμή όπου είχαν παρατηρηθεί πολύ θετικές εξελίξεις και ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση σχέση με το παρελθόν το απόθεμα του Μπακαλιάρου και του Σολομού. Δεύτερον, Ε, διάφορα ε, σκάφη εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση καταχώρησης των αλλιευμάτων ε, συγκεκριμένα όσα σκάφη είναι ε, κάτω των 8 μέτρων και ε, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία όταν υπάρχουν τέτοιε εξαιρέσεις δεν είναι πλήρη ούτε αξιόπιστα. Άλλα μέτρα, η χρήση των παρασυρώμενων δικτυών για την αλληλεία Σολομού επί τη βάση ενός ασφαλμένου επιχειρήματος ισχυρίζονται ε, κάποιοι ότι ε, επηρεάζονται και άλλα θαλάσσια είδη από την ε, αλία του Σολομού με δίχτυα. Αυτό δεν ισχύει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να εξετάσει περαιτέρω ε, ε, ε, αρνήθηκε συγγνώμη, να εξετάσει την επιρροή της χρήσης των σειρώμενων δικτύων για την αλία του Σολομού επί άλλων ειδών. Αυτά γίνανε το 2007. Αναφέρθηκα σε κάποια παραδείγματα αυτή τη παθογένεια του συστήματο που παρατηρείται στην περιοχή τη Βαλτική. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει αν ήταν περιφερειακή η διαχείριση των αλλιευμάτων ακόμη και αν ε, ε, καταφέρουμε να εφαρμόσουμε αυτή την αρχή της ε, περιφερειοποίησης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παρόλα αυτά δεν θα μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε κάποιες από αυτές τις απώλειες. Επίσης, απαξιώθηκε τρόπον την η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχασε την αξιοπιστία της, διότι ε, ο κλάδος κρίνει ότι είναι ανεύθυνη αυτή η δράση της Επιτροπής ε, που ε, υποχρεώνει, στριμώχνει τις χώρες της Βαλτικής να υποταχθούν ενώπιον της γραφειοκρατίας και Συνεχίζονται τα προβλήματα σε σχέση με την συλλογή και την, ε, ε, την ε, συλλογή και τη διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων. Παρατηρούνται αυτά τα προβλήματα ακόμη και σήμερα στις χώρες της Βαλτικής. Πιστεύω ότι εάν είχε προσφερθεί ε, στις χώρες της Βαλτικής ε, η δυνατότητα να διαχειριστούν ναι, τα αλλιευτικά τους αποθέματα και την ποσόστοση που έχουν ως προς τις αλλιευτικές ικανότητες θα ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση σίγουρα καλύτερη από ότι όταν λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις ε, στις Βρυξέλλες. Για να κλείσω θα αναφερθώ μόνο σε ένα εγγραφό που περιέχει όλα τα πετούμενα στοιχεία τα οποία ε, ε, στοιχειοθετούν αυτές τις ε, παρατυπίες που μόλις σας περιέγραψα. Θα διαβιβάσουμε το έγγραφο αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να συμβάλλουμε στην μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής βασιζόμενη στην επιστημονική ακρίβεια και αξιοπιστία και όχι στην άγρια φαντασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημιούργησε όλες αυτές τις παθογένειες στη Βαλτική. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Στίβενσον, ε, σας ευχαριστούμε κύριε Σόμπορκ. Ευχαριστώ. Ε, υπερβήκατε κατά τι το χρόνο αγόρευσης και σας ευχαριστούμε. Ε, πρα, παρακαλώ όλους τους ομιλητές να μην υπερβαίνουν τα 10 λεπτά. Ο Μπρέν, Ορίεν, ο γραμματέας ε, της ε, Ιρλανδικής Ένωσης των Επαγγελματιών του Κλάδου, ο πλευράς της θα πάρει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή Αλίας που μου επιτρέπει να θέσω υπόψη σας ορισμένα θέματα της μικρής κλίμακας αλίας. Όλοι νομίζω συμφωνούν ότι η περιφερειοποίηση είναι η καλύτερη δυνατότητα ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, εφόσον βέβαια υπάρχει η πολιτική βούληση και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο των χωρών μελών, να αντιμετωπιστούν δηλαδή οι περιορισμοί της συνθήκης της Λισαβόνας. Η μικρή κλίμακα παίζει σημαντικό ρόλο μέσα στην περιφερειακή κοινή αλληλευτική πολιτική, όπως και αν αυτή ε, οριστεί και όπως και αν επιτευχθεί. Διότι η μικρή κλίμακα αλληλεία είναι σημαντικός παράγοντας και για την απασχόληση και για την διατροφή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η στόλη της μικρής ε, κλίμακας αλληλείας, λιγότερο από 12 μέτρα δηλαδή, είναι 40%, ανέρχονται σε 40% της απασχολήσεως και 80% των σκαφών. Αν και από άποψη μικρού τονάζ και ε, συνολικών υποδυνάμεων είναι πολύ μικρότερη. Χωρίς να λάβουμε καν υπόψη τις παρελκόμενες ε, θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Η αλία μικρής, κλίμακα είναι στρατηγικά σημαντικός παράγοντας στο ευρωπαϊκό ενωσιακό επίπεδο από κοινωνικο-οικονομική σκοπιά και κυρίω για τι πιο περιοχέ τη Ευρώπη, όπου αν εξαφανιστούν οι αλίες αυτέ θα έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στην απασχόληση. Παίζουν και σημαντικό ρόλο για την παροχή εναλλακτικών πηγών ε, για να παράγουν δηλαδή φρέσκο ψάρι για τοπικές και εξειδικευμένες αγορές μέσα σε μια προσπάθεια να φτάσουμε σε μια πράσινη οικονομία. Το ICSF θεωρεί ότι στην Ευρώπη οι μικρές κλίμακας αλλίες αποτελούν ένα σημαντικό υποτομέα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ειδικά μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή ελευτικής πολιτικής και γι' αυτό χαιρόμαστε που οι, Ευρω... οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται στην σημασία αυτή για τον νέο κανονισμό και για το νέο Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, το EMFF. Θεωρούμε ωστόσο ότι αυτές οι προτάσεις πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο και χρειάζεται περισσότερη συνοχή ανάμεσα στις διάφορες διατάξεις, γιατί έχουν μεγάλη σημασία για τις μικρής κλίμακας αλίας. Για παράδειγμα, η πρόταση για τις μεταβιβάσιμες αλλιευτικές παραχωρήσεις έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την θέση των μικρής κλίμακας ε, αλίας. Οι μεταφερόμενες παραχωρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ε, μεγαλύτερους ομίλους επιχειρήσεων και αυτό θα είναι άσχημο για τις μικρές και ε, μικρές κλίμακας αλίας. Η μεσογειακή πλατφόρμα βιοτεχνών ψαράδων με συμμετοχή ψαράδων από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα έχουν τονίσει ότι η απαγόρευση των απορρίψεων θα οδηγήσει στην ε, αλία και εκφόρτωση ανώριμων ψαριών και αυτό θα είναι ε, κάτι το οποίο θα ευνοήσει τελικά τις ε, απορρίψεις. Οι σχετικές διατάξεις είναι καλύτερα να ληφθούν στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ανατομέα αλίας μέσα σε ένα πλαίσιο που θα θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με γενικούς στόχους για μείωση των, της ικανότητα. ικανότητας. Ποιοι είναι οι παράγοντες εν προκειμένου, ποιοι είναι οι φορείς, για ποιους μιλάμε. Όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι μικρές κλίμακας αλίες στην Ευρώπη έχουν εξελιχθεί μέσα στον χρόνο και στον χώρο από συγκεκριμένα οικολογικά και κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά πλαίσια και έχουν μάλλον διαχαρακτηρίζονται από διαφοροποίηση. Οποιαδήποτε λοιπόν συζήτηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι εδώ υπάρχει και ένας, μια πρόκληση σχετικά με τον ορισμό. Οι ορισμοί δεν μπορούν να εφαρμόζονται συνολικά. Κάτι που μπορεί να είναι μικρή κλίμακα σε μία κατάσταση μπορεί να είναι μεσαία ή μεγάλη κλίμακα αλλού. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον ορισμό των μικρή κλίμακα αλλιών. Και αυτό οφείλει να ληφθεί υπόψη, καθώ επίση και η ανομοιογένεια των μικρή κλίμακα αλλιών. Μιλούμε για τους πλειοκτήτες και τα πληρώματα μικρών σκαφών που χρησιμοποιούν αλληλευτικά εργαλεία μη ελκόμενα, δηλαδή στατικά, και που ε, δραστηριοποιούνται στους τοπικούς τους ψαρότοπους. Και μέσα σε όλη την αλυσίδα της αλίας πρέπει να είναι μικροί οι φορείς, δηλαδή ε, με τις συζύγους οι οποίες συνεργάζονται με μικρές άλλες επιχειρήσεις, των οποίων το καθεστώς οφείλει να αναγνωριστεί. Επίσης, οι εργάτες που διορθώνουν τα δίχτυα, ή όπως στην Ισπανία είναι οι γυναίκες που το κάνουν αυτό, οι μικρής κλίμακας μεταποιητές και οι αντιπρόσωποι αυτών των φορέων. Ωστόσο, μικρή κλίμακα, όπως και αν οριστεί η αλία της μικρής κλίμακας, θα πρέπει να είναι λειτουργική. Ο ορισμός που μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασισμένος στο μήκος του σκάφους και στα αλλιευτικά εργαλεία νομίζουμε ότι είναι πολύ περιορισμένος και δεν λαμβάνει υπόψη της, την ανομοιογένεια των διαφόρων αλλιών ε, τοπικά. Ναι μεν θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά αυτός οφείλει να λάβει περισσότερο υπόψη τις τοπικές ανομοιογένειες και με κάποια ευκαμψία, να επιτρέψει δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη και τοπικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες με τρόπο που να είναι λογικός. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει κάποια ευκαμψία σε ό,τι αφορά το μήκο του σκάφου και τον αλληλευτικό εξοπλισμό, να λαμβάνει υπόψη την χωρητικότητα ή τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται και ε, ελκόμενα αλληλευτικά εργαλεία. Σε πολλά μέρη της Ευρώπης οι αλληλείς έχουν λάβει, λαμβάνουν μέρος και σε μια προσπάθεια θέσπισης των βέλτιστων πρακτικών. Αυτές οι πρωτοβουλίες μάλιστα είναι πολύ καλά θεμελιωμένες, τεκμηριωμένες. Αυτά γίνονται κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και στο περιφερειακό επίπεδο και να γίνουν σεβαστά από τους κανονισμούς και τα νομοθετικά πλαίσια που επεξεργάζεται το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό λοιπόν οι τοπικοί παράγοντες να συμμετάσχουν στις περιφερειακές αυτές εξελίξεις και να μπορέσουν να εκφράσουν απόψεις μέσω των αρμόδιων συμβουλευτικών οργάνων. Πώς θα συμμετάσχουν λοιπόν οι τοπικοί φορείς στην περιφερειοποίηση για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εκεί αντιμετωπίζουν πολλούς περιορισμούς και μειονεκτήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη διάρκεια της περιφερειοποίησης όπως για παράδειγμα πολλές, πολύ μικροί ψαράδες δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένες οργανώσεις η ε, σωματεία και δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Άλλες οργανώσεις στις οποίες ανήκουν συχνά δεν είναι ενσωματωμένες σε, για παράδειγμα, οργανώσεις παραγωγών ή ε, συνδικάτα τα οποία να είναι αναγνωρισμένα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όταν ανήκουν σε τέτοιους φορείς, συχνά τα συμφέροντά τους παραβλέπονται λόγω του ότι η οργάνωση είναι τέτοια που δεν τα λαμβάνει υπόψη. Οι... Δεν εκπροσωπούνται επαρκώς οι μικροί ψαράδες ούτε στα αρμόδια όργανα. Χρειάζονται λοιπόν οργανισμοί οι οποίοι θα απηχούν συγκεκριμένα τα συμφέροντα των μικρών ψάραδων, της μικρής κλίμακας, των μικρών κλίμακας αλλιών που θα πρέπει επίση να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Να έχουν το δικαίωμα δηλαδή ανάληψης πρωτοβουλίας. Η περιφερειοποίηση οφείλει να λάβει υπόψη και μηχανισμούς που να επιτρέπουν και άνωθεν και κάτωθεν την κίνηση αυτή. Ένα παράδειγμα ίσως είναι αυτό που δίνει η Μεσογειακή Πλατφόρμα Βιοτεχνών Ψαράδων που προτείνει σχέδια συνδιαχείρισης από επιτροπές συνδιαχείρισης που θα δίνουν τη δυνατότητα να συμμετάσχει να συμμετάσχουν οι τοπικοί ψαράδες με τη γνώση τους στην ε, επιστημονική ε, έρευνα και θεμελίωση. Αυτό μπορεί να περιλάβει μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης, ειδικά για ορισμένες περιφερειές και ορισμένες περιοχές, με επιτροπές συνδιαχείρισης, στις οποίες να συμμετάσχουν ντόπιοι ψαράδες, επιστήμονες και ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Να παρακολουθούν δε τα σχέδια διαχείρισης με μια βάση προσαρμογής. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν σχετικοί μηχανισμοί όπου τέτοιες προτάσεις να μπορούν να συζητηθούν, να έχουν επεξεργασία και να συμφωνηθούν. Βλέπω ότι λίγο ο χρόνος μου σιγά σιγά. Θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα να πω ακόμη ότι λίγη πρόοδος μπορεί να γίνει προς την κατεύθυνση του στόχου μας των βιώσιμων ε, αλλιών όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη μέσα στα, πλαίσια, στα συστήματα ε, ελέγχου. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα σύστημα διαχείρισης βασισμένο σε μια διαδραστική διαχείριση στη βάση της περιφερειοποίησης. Χρειάζεται λοιπόν μια διαδραστική προσέγγιση σε τρία επίπεδα. Το πρώτο που θα περιλαμβάνει τον τοπικό εντοπισμό προβλημάτων. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο της διαχείρισης. Το δεύτερο επίπεδο των ευθυνών θα είναι σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που θα έχει σχέση με τις θεσμικές διαδικασίες και την επίλυση διαφορών και ούτε Και το τρίτο επίπεδο, μετακρατικό δηλαδή, θα είναι η θέσπιση των κριτηρίων της ε, πολιτικής αυτής. Έληξε ο χρόνος μου και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριόρνταν και σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρόνο. Ελπίζω να μπόρεσαν και οι διερμηνείς να αποδώσουν τις ε, ιδιαιτερότητες ε, της ομιλίας σας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Χωσέ Μανώλη Σομπρίνο Ερέντια, ο οποίος είναι καθηγητής Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κορούνια στην Ισπανία. Καλησπέρα σας. Ε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω που καλέσατε έναν ακαδημαϊκό για να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση σχετικά με την ε, περιφερειοποίηση ή την αποκέντρωση της κοινής πολιτικής. Η την αποκεντρωση της κινησιλευτικης πολιτικης η προσεγγιση που θα κάνω εγώ στο ζήτημα της περιφερειοποίησης ε, θα είναι νομική η ευκαιρία δίνεται από την αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής που επιτρέπει για μια ακόμη φορά να αναρωτηθούμε αν ε, το ε, μοντέλο διαχείρισης ε, της ελευθερικής πολιτικής είναι το κατάλληλο ή αν θα προέκυπταν ε, ωφέλη για την ελευθερική διακυβέρνηση αν εισαγάγουμε νέα στοιχεία αποκέντρωσης και περιφερειοποίησης. Σε πολλά έγγραφα λέγεται ότι μια αποτελεσματική διαχείριση των ελευθερικών πόρων πριν από την αποκέντρωση Δηλαδή, ε, θεωρώντας ότι το σημερινό σύστημα έχει το μειονέκτημα να καλύπτει ένα υπερβολικά μεγάλο γεωγραφικό χώρο. Και ε, να εξηγιανθεί αυτό θα ήταν να πάμε προς ε, μία διαχείριση αναζώνησης της κινησιλευτικής πολιτικής που εμπνέεται ε, από την αρχή της επικορικότητας ή βάση κριτηρίων περιφερειοποίησης ή αποκέντρωσης. Αυτό το νέο μοντέλο θα ευνοούσε μια δημόσια διαχείριση πιο αποτελεσματική και διαφανή σύμφωνα με την καλή διακυβέρνηση που διακηρύσει η ίδια η πρόταση κανονισμού της Κομισιόν ε, στα εκτιμώντας 10 ε, και στο, άρθρο, στο 10 και στο άρθρο 4. Όμως ε, η αποκέντρωση και η περιφεροποίηση απαιτεί καταρχήν να πάμε πιο πέρα από τα σημερινά περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Είναι απλώς γνωμοδοτικά και να δημιουργηθούν νέε περιφερειακές επιτροπές διαχείρισης που θα αποτελούνται από τα κράτη-μέλη που θα είχαν ένα πραγματικό ενδιαφέρον ε, για ε, τα ελεύματα μια συγκεκριμένη ζώνη ή ενός τρόπου αλίας δίνοντας αυτές επιτροπές δυνατότητα να συμμετέχουν έχουν απευθεία στις νομοθετικές διαδικασίες. Με αυτό θα δινόταν περιεχόμενο πραγματικό στι προτάσει περιφερειοποίηση τη κοινή ελευθερική πολιτική, ε, χωρί να πέφτουμε στην επανεθνικοποίηση αυτή. Για ε, να αναπτύξω αυτή την ιδέα. Καταρχήν θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω κάποιες έννοιες που χρησιμοποιούνται, κατά κατόπιν να τονίσω ε, ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι, τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται και κατά κατόπιν να προσδιορίσω τις διάφορες διαδικασίες που επιτρέπουν σε αυτούς τους πρωταγωνιστές να έχουν ε, συμμετοχή στην νομοθετική διαδικασία. Καταρχήν, ε, η ορολογία. Το πρώτο που επιστά την προσοχή ενός ακαδημαϊκού αν μελετήσει τα διάφορα έγγραφα ε, των διάφορων οργάνων και θεσμών ε, σε σχέση με την αναθεώρηση της κινησιλευτικής πολιτικής ε, είναι ότι χρησιμοποιείται μία σειρά όρων και δεν υπάρχει ακρίβεια. Χρησιμοποιούνται σαν να επρόκειτο για όρους συνώνυμους ενώ δεν είναι περιφερειοποίηση, αποκέντρωση Μιλάμε επίσης για επικουρικότητα. Γι' αυτό θεώρησα ότι είναι σκόπιμο να παρουσιάσω τρεις σύντομες ιδέες για να διαφοροποιήσω της ενίσευτες Διακυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μια μορφή διαχείρισης ε, όπου δεν έχουμε μια μεμονωμένη δράση μιας πολιτικοδικητικής ελίτ, ε, ομογενοποιημένης και κεντρικής, αλλά υιοθετούνται μορφές διαχείρισης σε διάφορα επίπεδα. Συνοδεύεται από επίθετα ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, παγκόσμια διακυβέρνηση, διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα κτλ. Και στα έγγραφα βλέπουμε τη χρήση σε διάφορες, ε, των όρων αυτών σε διάφορε στιγμέ, Αν ε, θέσουμε τη διακυβέρνηση στο ιστορικό τη κοινή ελευθερικής πολιτική, αυτό θα σημαίνει ότι το πολιτικό ευρωπαϊκό παιχνίδι θα έπρεπε να αναπτυχθεί σε πολλαπλό επίπεδα και ότι οι δημόσιε διοικήσει, οι ευρωπαϊκέ, οι εθνικέ, περιφερειακέ και τοπικέ, αν και διατηρώντα την ηγετική θέση στην πρόταση των, των δημοσίων πολιτικών, θα έπρεπε να τι ανοίξουν στου ε, κύριου πρωταγωνιστέ τη κοινωνία των πολιτών. Επίσης γίνεται λόγος για επικουρικότητα, αλλά επικουρικότητα είναι κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για μια αριθμιστική αρχή του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το οποίο η Ένωση, εκτός από τις περιπτώσει που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, παρεμβαίνει μόνο στο βαθμό που η δράση είναι πιο αποτελεσματική από την παρέμβαση σε ε, άλλα επίπεδα. Δεδομένου ότι η προστασία των διατήρηση των πόρων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή να μιλάμε για την χρήση της αρχής της επικουρικότητας. Ε, ναι, για άλλου ε, τομεί τη ε, κοινή ελευθερική πολιτική, αλλά και του πόρου. Αποκέντρωση. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για την δράση μεταφορά ορισμένων ιδιωτήτων από την κεντρική διοίκηση σε κάποιε ενδιάμεσε διοικήσει, τι οποίε αναγνωρίζεται αυτονομία για την διαχείριση το συμφερόντων του. Η είναι ένα ακόμα βήμα παραπέρα, ε, γιατί ε, πέρα από τις... Ε, έχουμε μάλλον τις νομοθετικές προτεραιότητες, αρμοδιότητες ή περιοχές θα έχουν τέτοιες νομοθετικές προτεραιότητες ε, ή τα όργανα μάλλον μέσω των οποίων ασκούν νομοθετική δράση περιφερειακές θα πρέπει να καθορίσουμε τι θεωρούμε περιφέρεια, τι είναι περιφέρεια για την κοινή ελευτική πολιτική θα μπορούσε να οριστεί ε, είτε λόγω της θαλάσσιας πολιτικής είτε λόγω ε, συγκεκριμένου είδους αλίευσης και ε, το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να έχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον σε αυτό το είδος αλίας και έχουμε και ε, την μεταφορά των αρμοδιοτήτων από ένα ανώτερο ιεραρχικά όργανο σε ένα όργανο που είναι ιεραρχικά κατώτερο αλλά μέσα στην ίδια δημοσία διοίκηση. Εκεί έχουμε γεωγραφική αποκέντρωση, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο, μιλάμε για την ίδια δίκηση. Δηλαδή, αυτό ε, τι θέλει να κάνει τώρα ε, η κοινή αλληλευτική πολιτική. Θέλει να προβεί σε ποιο είδος αποκέντρωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τους πρωταγωνιστές, που είναι το δεύτερο μέρος, νομίζω ότι η διαδικασία της αποκέντρωσης υπερφυροποίησης απαιτεί μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών όλων των ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια της, του σχεδιασμού και της εφαρμογής ε, της κινησιδευτικής πολιτικής, αλλά δεν εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερομένοι με τον ίδιο τρόπο σε όλη την ε, κάλπ και ιδίω ό,τι αφορά τις ε, διάφορες ε, θαλάσσιες λεκάνες και στα διάφορα είδη αλίας. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν συγκεκριμένο ενδιαφέρον και αν αυτό το δεκτούμε θα έπρεπε να ανοίξει ο δός για να επιτρεπεί μια ενισχυμένη συνεργασία που θα καθορίζεται περιφερειακά. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα όργανο, ένα είδος μίνι κορεπέρ ή μια ομάδα εργασίας που θα υποκαλούσαμε Επιτροπή Περιφερειακής Διαχείρισης ε, που θα λειτουργούσε βάση ε, και των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων που θα είχαν περισσότερες αρμοδιότητες. Ό,τι αφορά τον θα έπρεπε να συμπίπτει με τις ε, Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές. Εκεί θα έπρεπε να εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον, αλλά επίσης και οποιοδήποτε κράτος μέλος που το επιθυμεί, που θα μπορούσε προσωρινά ή μόνιμα να αποτελεί μέλος πλήρους δικαίου. Επίσης, σε αυτές τις επιτροπές θα συμμετείχε και εκπρόσωπος κομισιών ε, που θα μπορούσε να έρθει λόγο, αλλά χωρίς ψήφο. Σε σχέση με τη λειτουργία, θα λειτουργούσε η επιτροπή αυτή αυτόνομα βάσει πρόταση της κομισιών ή κατόπιν αιτήματο του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ή κάθε φορά που θα χρειαζόταν η υιοθέτηση κάποιας απόφασης. Η απόφαση θα λαμβανόταν με την μορφή γνωμοδότησης, πριν από την υιοθέτηση της γνωμοδότησης, ε, κάθε επιτροπή θα έπρεπε να λαμβάνει κάποιες εκθέσεις ε, που θα μπορούσαν να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα σε σχέση με τα θέματα που θα συζητούνται στο Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, ε, από το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, από την Επιτροπή των Περιφερειών. Σε ό,τι αφορά τώρα την συμμετοχή στι νομοθετικέ διαδικασίε, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μια γενική διαδικασία και μια ειδική διαδικασία γενική διαδικασία θα έπρεπε να κάνουμε μια διάκριση ανάλογα ε, με το αν η απόφαση μόνο από το Συμβούλιο, η Επιτροπή η Περιφερειακή θετούσε μια γνωμοδότηση βάση της πλειοψηφίας όπως λέγεται στο ε, άρθρο 238 και θα διαβιβαζόταν ως σημείο α στο Συμβούλιο και κατόπιν θα ακολουθούνταν η κανονική διαδικασία, η τακτική διαδικασία λειτουργία της ΚΟΡΕΠΕΡ και του Συμβουλίου αν ε, πρόκειται για θέματα που πρέπει να ακολουθήσουν ε, την τακτική νομική διαδικασία, εδώ ε, θα είχαμε κάτι παρόμοιο από το Οικονομικό Κοινωνικό Συμβούλιο και με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάλληλη στιγμή. Η ειδική διαδικασία θα θεσπιζόταν για την περίπτωση που τα πολιετή σχέδια ε, που έχουμε πολιτεί σχέδια δίνοντας ε, τη δυνατότητα στο Συμβούλιο, μάλλον στην Επιτροπή Περιφερειακή Διαχείρισης να υιοθετήσει μέτρα που θα προσδιορίζουν τα μέτρα διατήρηση σχετικά με τα, τα μέτρα διαχείριση, τα μέτρα σχετικά με τα σκάφη κτλ. Τέλος, η μεταρρύθμιση της κοινή πολιτικής Πολιτική αντιμετωπίζει την πρόκληση να προσαρμόσει το σύστημά τη με στόχο να συνδυάσει αποτελεσματικά τη γενική εκπροσώπηση Ευρωπαϊκή Ένωση με την εδαφική εκπροσώπηση κράτη και περιφέρειες, δίνοντας και χώρο στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Αλλά αν ε, επιθυμούμε την περιφερειοποίηση θα πρέπει να καθορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο περιφέρεια και πώς τα κράτη-μέλη εμπλέκονται μέσα σε κάθε μία από αυτές τις περιφέρειες. Έτσι, μαζί με τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια που σήμερα ε, έχουν γνωμοδοτική λειτουργία θα έπρεπε να δημιουργηθούν και αυτές οι επιτροπές, περιφερειακές επιτροπές διαχείρισης που θα έπρεπε να συμμετέχουν στις νομοθετικές διαδικασίες φυσικά μέσα στα νομικά όρια που θεσπίζει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, professor. Σας ευχαριστούμε, Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ο επόμενος ομιλήτης, ο προτελευταίος αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος ε, Χουάν Μανουέλ Τρογίλο Καστήλιο, που είναι ο πρόεδρος ε, της ε, Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών και της Αλίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής καλησπέρα σα καταρχήν. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που καλέσατε την ETF για να εκφράσει την άποψή τη για το θεμελιώδες ε, θέμα της περιφερειοποίησης, της πολιτικής, ε, της κοινή πολιτικής και ιδίως ε, με στόχο να γίνουμε πρωταγωνιστές ε, λέγομαι χωάν Μανώλη Τρουχίγιο, είμαι πρόεδρος ε, της ε, ETF. ETF σημαίνει Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών. Μια συνδικαλιστική ομοσπονδία με 341 συνδικάτα που εκπροσωπεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους από τον τομέα της αλλιές και των μεταφορών από 41 χώρες. Εμείς εκπροσωπούμε το ε, συμφέρον των ε, μισθωτών ελαίων. Από την αρχή τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΛΠ, η περιφερειοποίηση παρουσιάστηκε και καλωσορίστηκε από τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη ω μία από τι πιο καινοτόμε πτυχέ που θα έπρεπε να παρουσιαστούν από τη μεταρρύθμιση αυτό οφείλεται επειδή ε, θεωρείται ως ένας ε, λογικός τρόπος ε, για να δοθεί αρμοδιότητα λήψη αποφάσεων όσο πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες και να παρακολουθούν την εφαρμογή. Σε αυτό το στάδιο παρόλα αυτά είναι δύσκολο να κρίνουμε πώς η περιφερειοποίηση θα είχε αντίκτυπο στην διακυβέρνηση της Αλίας καθώς η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό δεν είναι πολύ λεπτομερής. Η περιφερειοποίηση παραμένει αυτή τη στιγμή μια ιδέα παρά ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ε, αν στην αρχή της συζήτησης προβλεπόταν ε, να δοθεί ρόλος λήψη αποφάσεων στα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια και να διευρυνθεί η συμμετοχή τους ε, στα κράτη-μέλη, ε, η συμμετοχή των κρατών σε αυτά. Είδαμε στη συνέχεια ότι η διεύρυνση των ε, ΡΑΚ δεν θα σεβόταν τη συνθήκη και ότι η περιφερειοποίηση θα ήταν πολύ πιο περιορισμένη από ό,τι είχε προβληθεί αν και ακόμη δεν είναι πολύ σαφές ο τρόπος με τον οποίο η έννοια της περιφερειοποίησης θα εφαρμοστεί στην πράξη, ε, τη γνώμη μας, η περιφερειοποίηση, η αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων θα πρέπει να περάσει από μία ε, πολύ προσεκτική αξιολόγηση, όχι μόνο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της παροχής συμβουλών, αλλά και των ε, πρωταγωνιστών που θα συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και με το πώς θα το ανεπίσημο έγγραφο για την περιφερειοποίηση που πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, μας διαφωτίζει πολύ για τη μεταρρύθμιση και για τους ενδιαφερομένους που θα έπρεπε να εμπλακούν από τα κράτη-μέλη. Γιατί αναφέρεται γενικά στους αλείς, ε, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στις περιφερειακές επιτροπές. Έτσι λοιπόν, καταρχήν η διαδικασία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το σημείο αυτό τα περιφερειακά συμβούλια, τα γνωμοδοτικά συμβούλια θα μπορούν να παρέχουν συμβουλές στη διαδικασία. Αν όχι, θα έπρεπε να προσδιοριστεί ποιοι είναι οι υπόλοιποι που θα συμμετάσχουν, έχοντας κατά νου ότι γενικά τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια θα ε, πρέπει να σχεδιαστούν για να συμμετέχουν εκεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει να εγγυώνται ένα μηχανισμό ισορροπίας για να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους για μας είναι θεμελιώδες οι εργαζόμενοι μέσα από τα συνδικάτα τους να διαδραματίζουν ένα πρωταρχικό ρόλο στην διαβούλευση. Η ΤΥΦΗ e έχει την ε, πρόθεση να συνεχίσει να ασχολείται με το συντονισμό, ε, να συντονίσει του εργαζομένου στι περιφερειακέ επιτροπέ, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι πόροι και να διαβαστεί η φωνή όλων ε, των θυγόμενων εργαζομένων μέσω μια συγκεκριμένη γνωμοδοτική επιτροπή, αποφεύγοντα τον άχρηστο κατακαιρματισμό στην εκπροσώπηση των συμφερόντων. Σε ό,τι αφορά την, ε, τις επιτροπέ. επιτροπές. Θα πρέπει να διδαχτούν ε, οι επιτροπές αυτές από την εμπειρία των ΡΑΚ. η σύνθεση των συμβουλευτικών επιτροπών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα ε, με το σε ποια περιοχή εργάζεται κανείς. έτσι λοιπόν ε, τα ενδιαφερόμενα μέρη, η συμμετοχή ε, των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να διαφέρει. Σε κάποιο συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει ένα στάδιο αριθμό χωρών και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν θα και θα κανονίζετε το αριθμό των μελών ε, που θα συμμετέχουν στα διακυβερνητικά όργανα. Θα πρέπει επίση να υπάρχει εκπροσώπηση, να ελέγχεται εκπροσώπηση έτσι ώστε όσοι αποτελούν μέλη των ε, συμβουλευτικών οργάνων ή συμμετέχουν σε διαδικασία διαβούλευσης είναι πράγματι αντιπροσωπευτικοί και έχουν εντολή για να μιλήσουν εξ ονόματος συγκεκριμένης ε, ομάδας ενδιαφέροντος και ε, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, σε ορισμένα κράτη-μέλη η εκπροσώπηση των συμφερόντων ε, δεν είναι πολύ καλή. Η συνεργασία με τις εθνικές διοικήσεις θα πρέπει να καθορίζεται το συντομότερο δυνατόν ε, προκειμένου με αποτελεσματικό τρόπο να διατηρείται η ικανότητα δημιουργίας και έτσι λοιπόν θα πρέπει ε, οι πόροι να διατίθενται και μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και για να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί που έχουν νόμιμα ενδιαφέροντα και συμφέροντα έχουν ε, την δυνατότητα να συμμετέχουν στη συμβουλευτική διαδικασία και να συνεισφέρουν ενεργά σε αυτήν μπορεί η συμμετοχή αυτή να κοστίζει πάρα πολύ για τα ενδιαφερόμενα μέρη, κυρίως όταν υπάρχουν κεντρικές οργανώσεις που πρέπει να εργαστούν για να συντονίσουν την άποψη των μελών τους. Έτσι λοιπόν ε, συμβολεύουμε μία, να δίνεται μία ενίσχυση παρόμοια με αυτή που δίνεται στα ε, μέλη της Επιτροπής Αλίας και Δετοκαλλιέργειας και αυτό επιτρέπει να γίνονται στορικές συζητήσεις, να προετοιμάζεται η συμμετοχή στις συμβουλευτικές διαδικασίες. Επίσης πιστεύουμε ότι ένα βήμα όπως ε, η Επιτροπή Ιδιωτοκαλλιέργειας και Αλίας πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό είναι το μοναδικό βήμα όπου τα κύρια τμήματα του κλάδου ε, από την παραγωγή, τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις ομάδες καταναλωτών και τις οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συναντηθούν για να συζητήσουν τα οριζόντια θέματα που ενδιαφέρουν την αλία και την ιδατοκαλλιέργεια. Θα περιορίσω την παρέμβασή μου στα σημεία αυτά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά ευχαρίστω να απαντήσω αν έχετε ερωτήσει αργότερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Και τώρα. Θα δώσουμε το λόγο στον επόμενο μιλητή, τον ε, κύριο Βίκτορ Περνέρο, που είναι πρόεδρος των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων ε, των Δυτικών ε, και Ανατολικών Ιδάτων και, και Νότιων Ιδάτων και θα παρουσιάσει, όπως είπαμε, την κοινή θέση όλων των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα παρουσιάσω τα δύο έγγραφα. Το ένα έχει συμφωνηθεί και το άλλο έχει με πέντε ε, ψήφους εξ ονόματος ε, των 7 ε, γνωμοδοτικών συμβουλίων θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση που έστειλε στα ΡΑΚ για να προσεγγίσουμε το θέμα ε, αυτό της περιφερειοποίησης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της μελλοντική κάλπη. Πολλοί από εσά ε, θα γνωρίζουν ότι σήμερα υπάρχουν 7 περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, 5 είναι περιφερειακά, Βαλτική, Βόρεια Θάλασσα, ε, Βόρεια και Δυτικά, Μεσόγειος και Νοτιοδυτικά είδατε ένα από αυτό μελετά τα πελαγικά είδη και άλλο εκπροσωπεί τον στόλο μακράς απόστασης. Ε, πολλά ρακ ε, δραστηριοποιούνται ε, πέρα από τα κοινοτικά ύδατα και γι' αυτό πρέπει να συμμετέχουν σε διεθνείς οργανώσεις, σε περιφερειακές οργανώσεις ελίας και να ε, δημιουργούν επαφές σε αυτή τη ζώνη επιρροής. Γι' αυτό αποτελεί τιμή για μένα να παρουσιάσω την ε, κοινή άποψη των 6 ρακ σε σχέση με την περιφερειοποίηση. Επίσης θα στείλω στη συνέχεια την αποκλίνουσα θέση του ρακ βελαγικών ειδών λόγω της ειδική κατάστασης στην οποία βρίσκεται σε σχέση με το θέμα αυτό πολλοί από τους ε, άλλους προέδρους του ΡΑΚ παρευρίσκονται ως παρατηρητές αυτήν αυτήν ακρόαση και θα είναι στη διάθεσή σας για να μπορούν να παρουσιάσουν τις αντίστοιχες θέσεις του κάθε ΡΑΚ αν χρειαστεί. Η πράσινη βίβλος της Κομισιόν ε, σχετικά με την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ αναγνωρίζει το ότι η σημερινή ΚΑΛΠ δεν ήταν επιτυχής τη στιγμή που προσεγγίσαμε το βάθ, το, την ουσία των διαρθρωτικών προβλημάτων ε, που αφορούν την Ευρωπαϊκή Έλλη. Έτσι λοιπόν η σημερινή ΚΑΛΠ δεν μπόρεσε να πετύχει μια βιώσιμη ελεία των ε, ε, ε, πληθυσμών από την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σκοπιά, και αναγνωρίζει ότι βελτιώθηκε η κατάσταση στην περίπτωση ορισμένων αποθεμάτων. Η ίδια η Κομισιόν αναγνώρισε ότι ένα από του κύριου λόγου αυτή τη ανεπάρκεια είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία λήψη αποφάσεων, που ιδιαίτερα κεντρική που εστιάζεται από τα πάνω προς τα κάτω με υπερβολική εξάρτηση στην μικροδιαχείριση από την πλευρά των ευρωπαϊκών οργάνων. Αντιμετωπίζουμε σήμερα μία μοναδική ευκαιρία για να τελειώσουμε με, δώσουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση που θα μπορούσαμε να πούμε δυσλειτουργική. Η λύση Παρ' αυτά απαιτεί όλοι να προσεγγίσουμε το πρόβλημα από κοινού και με έναν φιλόδοξο τρόπο. Είναι σαφές ότι οι κανόνες η φυστάμενη κανόνε ελέγχου δεν ήταν αποτελεσματική και ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μία πιο καθολική και συμμετοχική εστίαση. Είναι σαφέ επίση ότι είναι συμμετοχή, θα είναι συμμετοχή ε, απαραίτητη όλων των ενδιαφερομένων μέρων, ε, σεβόμενη την καλή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Η ιδέα να προσεγγίσουμε τι αποφάσει, τι βάσει, έτσι όπω λέγεται στην πρόταση του βασικού κανονισμού για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΛΠ, είναι το κλειδί για να ξεβρούμε λύσεις ε, διαχείρισης ε, που θα σέβονται τις ιδιαιτερότητες ε, των περιφερειών, των θαλάσσιων λεκανών ή των συγκεκριμένων ειδών αλίας. Ε, το ανεπίσημο έγγραφο διαβούλευσης της Κομισιόν για την Περιφερειοποίηση που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο με σύντομο τρόπο παρουσίαζε το μελλοντικό τρόπο των μελλοντικών οργανισμών διαχείρισης και τη δέσμευση των ε, Περιφερειακών Συμβουλίων στη διαδικασία διαχείρισης. Η γενική φύση του εγγράφου αυτού παρόλα αυτά δεν ε, θέλει να δώσει προτάσεις σε συγκεκριμένους ορισμούς ε, σε σχέση με το πώς θα επιτευχθεί η περιφερειοποίηση. Η κυρία μας πρόκληση είναι να καθορίσουμε μια διαδικασία που θα επιτρέπει να θέσουμε στην πράξη ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί τη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων μερών, κράτη-μέλη, όργανα, τις επιθεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ΡΑΚ, Περιφερειακά Οικονομικά Συμβούλια, των Επιστημόνων, των ΜΚΟ και άλλων ενδιαφερομένων μερών που θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για την εκπόνηση προτάσεων που να συνάδουν με τις γενικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από ε, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πετύχουμε, να έχουμε βιώσιμη αλία και καλή διαχείριση από τη δημιουργία του στα ΡΑΚ μετατράπηκαν σε ένα θεμελιώδες ε, βήμα για την ανταλλαγή απόψεων για στρατηγικά θέματα μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών σε περιφερειακό επίπεδο και με εστίαση που βασίζεται στα ίδια Τα ΡΑΚ ενίσχυσαν τη συνεργασία, το σεβασμό και την κατανόηση μεταξύ του ελευτικού κλάδου και άλλων ενδιαφερομένων και ε, απόδειξαν ότι είναι αποτελεσματικός μηχανισμός για να ενημερώνονται τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ανησυχίες τους και τις ε, απόψεις τους. Τα ΡΑΚ ε, εξελίχθηκαν λοιπόν για να μετατραπούν σε ένα βήμα συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων και ενδιαφερομένων μερών και αποτέλεσαν συναφές τμήμα πολλών ευρωπαϊκών σχεδίων. Παρ' όλα αυτά, όλα όσα επιτεύχθηκαν μέχρι τώρα δεν είναι παρά η αρχή ενός ταξιδιού και μας μένει ακόμα πολλής δρόμος. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε βάσει των επιτυχιών των ΡΑΚ, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε με σαφήνεια το ρόλο που θα δοθεί σε αυτά τα μελλοντικά περιφερειακά μα σε αυτά μελλοντικά γνωμοδοτικά συμβούλια, καθώς και να έχουμε και ένα ρελιστικό πλαίσιο χρηματοδοτικής στήριξης για τη λειτουργία τους. Και τέλος, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα 7 ΡΑΚ, τα σημερινά, αν ε, και ε, ιδρύθηκαν βάσει ενός κοινού νομοθετικού πλαισίου, ε, έχουν βασιστεί στην εθνική νομοθεσία για τη δημιουργία της και χρησιμοποιούν μια σειρά διαφορετικών μηχανισμών. Έτσι λοιπόν τα ράκα έχουν ε, μεμονωμένα χαρακτηριστικά και εξελίχθηκαν διαφορετικά προκειμένου να μπορέσουν να διαρματίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργίες τους και να εκπροσωπούν τις απόψεις των μελών τους. Αυτό επιτρέπει τα ΡΑΚ ε, να έχουν ε, πολλές διαφορετικές απόψεις, ακόμη και αν ε, προσεγγίζουν οριζόντια θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως συμβαίνει και με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ. Συνοπτικά, τα ΡΑΚ πιστεύουν ότι η μελλοντική επιτυχία των γνωμοδοτικών συμβουλίων εξαρτάται από το εξή. Οι πολιτικοί ηθήνοντε, τα εφερόμενα μέρη και οι ακαδημαϊκοί επιστήμονε να συνεργαστούν από κοινού για να πετύχουμε μία κοινή αλευτική πολιτική επαρκώ αποκεντρωμένη και σύμφωνη με του στόχου τη διαχείριση. Ποια είναι τα κοινά σημεία. Τα 7 ρακ που εκπροσωπώ εγώ σήμερα θα επιθυμούσαν να δουν τη συμπερίληψη των ακόλουθων κοινών στοιχείων στην ε, αναθεωρημένη ΚΑΛΠ. Ένα, μία διαδικασία λήψης αποφάσεων λιγότερο ε, συγκεντρωτική και πιο διαφανή με μία περιφερειακή διάσταση. Το περιφερειακό πλαίσιο είναι σημαντικό καθώς η αποκεντρωμένη εστίαση θα έπρεπε να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των ε, μεμονωμένων ε, ειδών αλίας. Οι ΤΑΡΑΚ αναγνωρίζουν ότι η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται ε, όχι μόνο από τις ε, ικανότητές τους ε, ή από την ποιότητα των γνωμοδοτήσεών τους, αλλά και από την αποδοχή και από τη βούληση να ακολουθήσουν τις απόψεις τους όσοι τις ακούν. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά των ΡΑΚ να ξέρουν πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα οργανώσει το μοντέλο διχείρισής τους. Βάσει όσων ε, αναφερθήκαν έξι ΡΑΚ, με ενθουσιασμό υποστηρίζουν μια κάλπη που είναι λιγότερο συγκεντρωτική ε, και θα βασίζεται η διαχείρισή της στα αποτελέσματα και να διασφαλίζει έναν ισότιμο ρόλο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, με διαφανή τρόπο σε συγκεκριμένο είδο αλεία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με κοινού στόχου και κοινά κριτήρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει να αναπτυχθούν στη συνέχεια από οργανισμού διαχείριση που θα έχουν δημιουργηθεί για να προσεγγίσουν συγκεκριμένα ζητήματα σε επίπεδο θαλασσιών λεκανών ε, ή ανά αλίευμα. Ε, ως εναλλακτική ο καθορισμός ενός ε, νέου πλαισίου λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή νομοθετικών μέτρων θα μπορούσε να είναι κάτι που θα εξεταζόταν. Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει να τεθεί σε λειτουργία μια καινοτόμως διαδικασία για να αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο αποκεντρωμένο για τη διαχείριση ε, λιμάτων που να περιλαμβάνει και να προσδιορίζει όλες τις γενικές έννοιες όπως παραδείγματο χάρη τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, την ελευτική ικανότητα και την οικοσυστημική προσέγγιση. Και το πιο σημαντικό που διαθέτει έναν ανάθεστο, είναι να διαθέτει έναν ανάθεστο μηχανισμό με ε, καλά προσδιορισμένο για την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης. Η αποκέντρωση δεν πρέπει να αποτελεί μεταφορά προς νέες πολύπλοκες δομές σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά να πετύχει μια πιο διαφανή εστίαση της λήψης αποφάσεων από μια περιφερειακή προοπτική. Έτσι, επίσης, για να λειτουργεί μια αποκεντρωμένη διαδικασία αποτελεσματικά, θα πρέπει από την αρχή να τεθεί σε λειτουργία μια επίσημη διαδικασία που να καθορίζει το ρόλο κάθε πρωταγωνιστή στη διαδικασία και ταυτόχρονα να επιτρέπει την ευελιξία έτσι ώστε κάθε οργανισμός διαχείρισης να αποφασίζει για τις εσωτερικές διαδικασίες του και τη λειτουργία του αν ξεκινήσουμε από την προπόθεση ότι τα μελλοντικά πολιετή σχέδια διαχείρισης θα, θα περιβληθεί σε αυτά μόνο μια γενική ένας γενικός ορισμός ε, των γενικών εργών και των στόχων ε, που θα υλοποιήσουν τα κοινοτικά όργανα, όπως παραδείγματος χάρη τεχνικά μέτρα, όπως ελάχιστα μεγέθη, ε, παγορευμένες ζώνες κτλ. Θα πρέπει αυτά με ολοκληρωμένο τρόπο να συμφωνούνται σε περιφερειακό επίπεδο και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών. Σαν ε, εξαίρεση, όσων υποθήκαν παραπάνω, το, ρακ, το πελαγικό ΡΑΚ θεωρεί ότι επειδή τα κύρια πελαγικά αποθέματα είναι εξόχως αποδημητικά και είναι εκμεταλλευόμενα κοινά με τρίτες, από κοινού με τρίτες χώρες, ο πελαγικός τομέας θεωρεί ότι θα, ή θα έπρεπε να αποκλειστεί από τον τομέα με τη διαδικασία της αποκέντρωσης θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο όργανο αποκεντρωμένο διαχείρισης που να αναλάβει τα πελαγικά είδη. Αυτή η οντότητα θα είχε ε, αρμοδιότητες κατανάθεση και ρητή εντολή για να διαπραγματευτεί με τρίτες χώρες, καθώς διαφορετικά θα προσθεθόταν ένα ακόμη γραφειοκρατικό στρώμα σε αυτό το πολύπλοκο μοντέλο διακυβέρνησης. Το πελαγικό ΡΑΚ επίσης αντιτίθεται απόλυτα στην διαχείριση των πελαγικών ειδών με ξεχωριστό τρόπο ή στην διαφοροποίησή τους ανά περιφερειακές ζώνες. Τα μελλοντικά ΡΑΚ θα πρέπει να έχουν ένα ενισχυμένο συμβουλευτικό ρόλο που θα καθορίζεται με σαφήνεια. Οι γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα και να υπερισχύουν έναντι μεμονωμένων γνωμοδοτήσεων. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς ε, τα γνωμοδοτικά συμβούλια, ε, στα γνωμοδοτικά συμβούλια συμμετέχουν πάρα πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και ε, εκδίδουν αιτιολογημένες απόψεις όπου αναφέρονται οι απόψεις όλων των μελών τους. Τα ΡΑΚ είναι οργανισμοί όπου συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων μερών που προωθεί το έργο σε συνεργασία μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν τον ελευτικό κλάδο και την ερασιτεχνική αλία, τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ και άλλες ομάδες ενδιαφερόντων που συμμετέχουν ως παρατηρητές ε, από τις εθνικές δικήσεις και από τον επιστημονικό κλάδο. Ο κύριος στόχος των ΡΑΚ εκφράζεται ε, μάλλον αν το κράσουμε με απλό τρόπο είναι να εκδίδονται γνωμοδοτήσεις που θα βασίζονται ε, σε αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα διαχείρισης ε, για ε, μια ζώνη όπου δραστηριοποιείται το ΡΑΚ για να διασφαλίσουμε ότι οι γνωμοδοτήσεις που εκδίδονται από τα ΡΑΚ αναγνωρίζονται επίσημα από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα κράτη-μέλη Όσοι η ενιαία φωνή των ενδιαφερομένων μερών, ο στόχος των ΡΑΚ είναι να πετύχει θέσεις στην ένεση πάντοτε όταν αυτό είναι δυνατό. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αντικατοπτρίζονται πάντοτε οι θέσεις οι μειονεκτικές και γι' αυτό πιστεύουμε ότι σε αιτιολογημένες ε, ε Νομοδοτήσει πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα από τα ευρωπαϊκά όργανα και να υπερισχύουν έναντι συνεισφορών που κατατίθονται από άτομα ή οργανώσεις. Συγκεκριμένα όταν παρουσιάζεται μία ενιαία συμφωνημένη θέση. Ε, με στόχο να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ Ιράκ και ευρωπαϊκών θεσμών είναι σημαντικό η Κομισιόν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τακτικά να στελούν τα σχόλιά τους ε, στα ΡΑΚ ε, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις που έχουν παρουσιαστεί. Τα σχόλια αυτά είναι ουσιαστικά για να βελτιωθεί η λειτουργία των σημερινών ΡΑΚ και των μελλοντικών περιφερειακών σε γνωμοδοτικών συμβουλίων και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αιτιολόγηση σε σχέση με τους λόγους που θα έχουν οδηγήσει στην απόφαση ε, να συμπεριληφθούν ή να απορριφθούν οι συστάσεις ε, των ΡΑΚ. Και τέλος, τα ΡΑΚ θα επιθυμούσαν ε, να ξεκαθαρίσει ο ρόλος των μελλοντικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και να καθοριστεί η συνεισφορά τους στα διάφορα είδη διαβουλεύσεων που προωθεί η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Αυτό θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει επίσης το βαθμό της έμφασης ή του βάρους που δίνεται στις γνωμοδοτήσεις των γνωμοδοτικών συμβουλίων στις εν λόγω Ανεξάρτητα από τη δομή ή το μοντέλο διαχείρισης που θα επιλεγεί, οι λειτουργίες και τα καθήκοντα των ε, γνωμοδικών συμβουλίων θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια στον κανονισμό της νέας κάλπ. Υπάρχουν ε, σαφή ωφέλη που προέρχονται ε, από ε, μία δομή τέτοια. Τα ΡΑΚ έχουν κάνει κάποιες προτάσεις σε σχέση με το πώς να βελτιωθεί η λειτουργία τους και η μεθοδολογία εργασίας και οι προτάσεις αυτές είναι διαθέσιμες ε, στα έγγραφα που παρουσιάζονται ως παράρτημα σε αυτή τη σημερινή ομιλία μου στα ε, γνωμοδοτικά συμβούλια σε πολλές περιπτώσεις έχουν ε, λειτουργήσει ως όργανα διαμεσολάβησης ε, τη στιγμή που υπάρχουν οξύνσεις μεταξύ των αλλιέων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς τα μελλοντικά γνωμοδοτικά συμβούλια θα μπορούσαν να πετύχουν γνωμοδοτήσεις βάσει αποδεικτικών στοιχείων και όταν είναι δυνατόν να υπάρχει και συνένεση για στρατηγικά ζητήματα. Ε, λοιπόν, αυτό το επίπεδο ολοκλήρωση είναι ουσιαστικό και μόνο θα επιτευχθεί αν υπάρχει σαφή κατανόηση τη λειτουργία των Γνωματικών Συμβουλίων και, ένας, ε, και έναν ορισμό και αναγνώριση ρητή του ρόλου τη. Πρέπει να διαχειριστούμε τι προσδοκίε όλων των μερών για αυτό το σημαντικό θέμα. Όμω, υπάρχει μια κοινή ευθύνη από την πλευρά τη Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και τα κράτη-μέλη για να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε περιορισμού είτε νομοθετικού είτε άλλη φύση, που θα μπορέσουν να θέσουν εμπόδιο στην πραγματική ανάπτυξη μιας περιφερειακή ε, διαχείριση ε, της Ελίας με πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Τα ΡΑΚ χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση για να βελτιώσουν την εσωτερική τους λειτουργία και να μπορούν να ολοκληρώσουν τις αυξημένες τους ευθύνες ασκώντας τα καθήκοντά του στα πλαίσια μια αναθερμένη κάλπη. Η αναγκαιότητα αύξηση τη χρηματοδότηση και απόκτηση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία θέθηκε από την ε, ομάδα ε, Interact στην Επιτροπή σε διάφορες περιπτώσεις, σε διάφορες συντονιστικές συνεδριάσει και με επιστολές. Τα ΡΑΚ θεμελίωσαν την αναγκαιότητα για ε, τέτοιο αίτημα στα συμπεράσματα που συμπεριλήφθησαν στην ανακοίνωση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της λειτουργία. Υγεία των ΡΑΚ δημοσιεύτηκε το 2008 και σε κατόπιν έκθεση ανεξάρτητων ε, ε, συμβούλων που δημοσιεύτηκε το 2010 οι οποίοι ζητούν ε, την πρόσθετη χρηματοδότηση για τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Στη βάση αυτή θα έπρεπε να αυξηθούν τα σημερινά επίπεδα χρηματοδότησης στο ΡΑΚ προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό τρόπο και να αναπτύσσουν δραστηριότητες πέρα από το σημερινό πλαίσιο που σήμερα, δράσεις τους που σήμερα περιορίζεται σε μία σειρά στρατηγικών δράσεων σε τήσια βάση τα ΡΑΚ. Πρέπει να έχουν την οικονομική ικανότητα και την δημοσιονομική ευελιξία για να μπορούν να αναλαμβάνουν δράση και από πριν. Προς αυτή την κατεύθυνση μια μεγαλύτερη ευελιξία σε γραμμές προπολογισμού θα επέτρεπε στα ΕΡΑΚ να είναι ικανά γρήγορα να προσαρμοστούν ε, σε μεταβαλλόμενες ε, περιστάσεις. Το μελλοντικό ταμείο θάλασσας και θα έπρεπε να επιτρέψει τη χρηματοδότηση διεθνικών σχεδίων από μια περιφερειακή βάση αντί να εξαρτάται από μεμονωμένα αιτήματα για κάθε ένα από τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται. Αυτό θα επέτρεπε στα μελλοντικά συμβουλευτικά, γνωμοδοτικά συμβούλια, με συγχωρείτε, να έχει πρόσβαση σε κοινά ε, project ε, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις. Έτσι λοιπόν τα ΡΑΚ προτείνουν ως ιδέα να διευνήσουν ότι το μελλοντικό ταμείο θα προβλέπει μια διαδικασία ταχείας οδού έτσι ώστε τα γνωμοδοτικά συμβούλια να μπορούν να ζητήσουν συγκεκριμένους πόρους για την ανάπτυξη ε, project που σχετίζονται άμεσα με τις ε, προτεραιότητες τους σχέδια διαχείριση, παραδείγματο χάρη, τεχνικά μέτρα, μείωση των απορρίψεων, η εξυγίανση, ε, αντιμετώπιση τη έλλειψη δεδομένων. Και, θα χρειαστεί στο βαθμό που θα χρειαστεί πολυετής σχεδιασμός των δραστηριοτήτων τους ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και τη δημοσιονομική ευελιξία, τα ΡΑΚ επίσης θα ήθελαν να συμμετάσχουν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων έρευνας αυτή η ολοκλήρωση θα υποστήριζε την ανάπτυξη μιας πιο στρατηγικής σχέσης και ε, μακροπρόθεσμα με την Κομισιόν μέσω της εναρμόνισης των προγραμμάτων, των πολιετών προγραμμάτων εργασίας των ΡΑΚ και πιο ευρεία έρευνα τη Κομισιόν. Θα έπρεπε να αναμένεται μια μεγαλύτερη συμμετοχή και δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών και των επιστημόνων ε, στο έργο των γνωμοδοτικών συμβουλίων και καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους. Η Κομισιόν θέσπισε ένα επίσημο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ΡΑΚ, του ΆΙΣΙΣ και της Οικονομικής Τεχνικής και Επιστημονικής Επιτροπής Αλίας που λειτουργεί επαρκώς. Έγιναν σημαντικές πρόοδοι ε, σε σχέση με ε, την αναθεώρηση των πολιετών ε, σχεδίων που ισχύουν. Στο βαθμό που προχωρά αυτό το έργο θα προκύψει και η απέτηση ε, να, να αναθεωρείται η γνωμοδότηση των επιστημόνων. Έτσι λοιπόν τα μελλοντικά ΡΑΚ θα πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στους επιστημονικούς πόρους προκειμένου να μπορέσουν να υποστηρίξουν τη διαδικασία αυτή με την έκδοση ε, γνωμοδοτήσεων είναι, είναι σημαντικό ε, θα, να ε, γίνει αυτό σε ένα έγκαιρο στάδιο έτσι ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στην εκπόνηση και ε, παραγωγή γνωμοδοτήσεων ε, γίνεται εκ των προτέρων ε, και σέβεται τις προτεραιότητες της Κομισιόν. Θα πρέπει ε, να, έτσι μάλλον θα ενισχυθεί η νομότητα των αποφάσεων συμπερασματικά. Η συμμετοχή και η δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών που εκπροσωπούνται στα ΡΑΚ θα πρέπει να συνεχιστεί ως σημαντική συνιστόσα της διακυβέρνησης σε επίπεδο του ΣΚΑΛΠ, όποια και αν είναι η μορφή που θα επιλεγεί για την υλοποίησή της. Η δουλειά των ΡΑΚ έχει εξελιχθεί σημαντικά από τη δημιουργία τους σύμφωνα με την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ. Καθ' όλα αυτά τα έτη παγιώθηκε η ικανότητα των ΡΑΚ ως βήμα ανταλλαγή απόψεων και μεταφοράς γνώσης. Θα θέλαμε αυτή η συμμετοχή να συνεχιστεί και στο μέλλον και ιδίω να δοθεί ένας ενισχυμένος ε, ρόλο και καλύτερα προσδιορισμένο στα ΡΑΚ. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι και υπαρκώς ευέλικτοι πόροι για να μπορέσουν ε, να ε, παρέχουν στους πολιτικά ηθήνοντες τις κατάλληλες συστάσεις. Η περιφερειοποίηση αποτελεί ταυτόχρονα μία πρόκληση σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή της και μία ευκαιρία για να αντικατοπτρίζεται η διαφοροποίηση των θαλασσών και των ευρωπαϊκών ελευτικών ειδών. Ε, και τώρα, αν μου επιτρέπετε, στο, μικρό, στο λίγο χρόνο που έχω, στα 7 λεπτά θα αναφέρω τις συγκεκριμένες ιδέες των διάφορων περιφερειακών ε, επιτροπών για το ΡΑΚ της Βαλτικής. Ε, το ΡΑΚ δεσμεύτηκε στο να έχει ένα ρόλο στην μελλοντική πολιτική για τη Βαλτική είναι πεπισμένο ότι η περιφερειοποίηση είναι μια αναγκαιότητα για τη μελλοντική κάλπε και δεσμεύτηκε να λειτουργήσει με πρακτικό τρόπο. Ο στόχο θα πρέπει να είναι να καταλήξει σε καλή υπεργοή με τη συμμετοχή ε, τη και το συντονισμό στην γλώσσα ε, περιοχή της Βαλτικής σε σχέση με άλλες περιοχές ε, ε, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση γιατί έχει συστηθεί το Baltfish. Το Baltfish πιστεύει ότι αποτελεί ένα βήμα προς τα μπρο στην κατάλληλη κατεύθυνση και θα ήθελε να αναπτυχθεί το βήμα Baltfish μέσα στο ίδιο το ράκ της Βαλτικής. Το Baltfish θα μπορούσε να λειτουργήσει ως όργανο εκπροσώπησης όλων των ενδιαφερομένων μερών, θα μπορούσε να προετοιμάσει συστάσεις της ε, περιοχής για τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα μπορούσε να συμφωνήσει για θέματα που έχουν να τοθεί ε, στη Βαλτική ή στα κράτη-μέλη της Βαλτικής. Το Baltic Sea Rack σήμερα διαπραγματεύεται με τα κράτη-μέλη της Βαλτικής στο πλαίσιο της επόμενης συνεδρίασης το Μάιο. Το Μάιο. Η περιφερειοποίηση θα είναι στην ατζέντα αυτής της συνεδρίασης. Έτσι λοιπόν από το ΡΑΚ της Βαλτικής υπάρχει ένα σαφές σχέδιο ανάπτυξης της περιφερειοποίησης μέσω του Baltfish το ρακ της Βόρειας Θάλασσας. Ε, τώρα, η άποψη αυτού του ρακ είναι ότι η εξάρτηση σε μία εστίαση ε, ελέγχου διαχείριση που να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη είναι ο πρώτος ρόλος για τον οποίο η ΚΑΛΠ ε, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Το επόμενο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό και πιο ευέλικτο και πιο απλό. Το ΡΑΚ της Βόρειας Θάλασσας υποστηρίζει μία ε, πραγματικά αποκεντρωμένη εστίαση θα πρέπει να καθοριστεί μια σειρά στόχων και αρχών ε, στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως οι λεπτομέρειες θα πρέπει να καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών μελών και στις περιφερειακές επιτροπές, σε μια περιφερειακή διαδικασία και διαφανή με την πλήρη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών. Αυτό θα οθήσει την αρχή της αυτοδιαχείρισης της Ελίας. Ε, το πιστεύει το μοντέλο αποκέντρωσης που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο αποτελεσματικό για τη διαχείριση της ελίας σε περιφερειακό επίπεδο στη Βόρεια Θάλασσα θα ήταν μια οντότητα που θα αναπτύσσει πολιτικές και θα επιβλέπει την εφαρμογή της νομοθεσίας στη Βόρεια Θάλασσα σύμφωνα με τους κανόνες, τις αρχές και τους στόχους που τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, το ΡΑΚ ε, μακρά απόσταση. Αυτό θεωρεί ότι μια ισορροπημένη εκπροσώπηση των ε, ομάδων συμφερόντων στα ΡΑΚ στι διαπραγματεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη-μέλη και με τι τρίτε χώρε θα μπορούσαν να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τη διαπραγμάτευση, συνεισφέροντα έτσι στον κύριο στόχο τη ΚΑΛΠ που είναι η προώθηση των αρχών τη υπεύθυνη και βιώσιμη αλληλεία, ελαχιστοποιώντα τον αντίκτυπο των πολιτικών ε, συμφερόντων. Έτσι, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΛΠ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να βρει ένα μηχανισμό που να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις αντιδράσει όλων των πρωταγωνιστών του ΡΑΚ Μακρά Απόσταση κατά τη διάρκεια τη διαπραγματεύση των συμφωνιών και στα πλαίσια των ΠΟΔΑ. Λοιπόν, ΡΑΚ Μεσογείου, περιφερειοποίηση. Η έλλειψη ενό ε, πλαισίου διακυβέρνηση περιφερειοποιημένη ε, ε, καθιστά πιο δύσκολη την μεταρρύθμιση που έχει προβλεφθεί για τα είδη της Μεσογείου και το ΡΑΚ της Μεσογείου πιστεύει ότι τα πολιτή σχέδια δράσης, αυτά καθ' αυτά, αποτελούν μια απάντηση στην απέτηση μιας προσαρμοσμένης διαχείρισης των ευρωπαϊκών θαλασσών και προτείνει να εξελιχθεί ε, η διαμόρφωσή τους, δηλαδή να συμμετέχουν περισσότερο τα ενδιαφερόμενα μέρη, τρακ του Νότου το ΡΑΚ αυτό προτείνει να τεθεί σε εφαρμογή ταχαίωση περιφερειοποίηση στη δική του ζώνη αρμοδιότητα μέσω της δημιουργίας ομάδων ε, σχεδιασμού για την εκπόνηση συγκεκριμένων ε, κανόνων. Οι ομάδες αυτές περιορισμένη σύνθεση, 10 ατόμων το πολύ θα ομαδοποιήσουν τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις και θα συμμετέχουν και επιστήμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Κάθε ομάδα ε, θα παρακολουθείται από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η μεθοδολογία εργασίας επιτρέπει τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί ε, τους διάφορους πρωταγωνιστές σε απόσταση και απλώς ε, τους υποβιβάζει σε οι συγκητές γνωμοδοτήσεων ε, θα μπορούσε διαφορετικά να υπάρχει μια οριζόντια συζήτηση που επιτρέπει και την ανάληψη κοινών δράσεων και αυτό θα αποτελεί εγγύηση καλύτερη εφαρμογή ε, και κατόπιν αποδοχή. Έτσι, η μέθοδο αυτή εγγυάται και την συνοχή και την κοινή χρησιμοποίηση των επιστημονικών και ανθρώπινων πόρων των διάφορων δομών. Προσπάθησα να σεβαστώ το χρόνο, Πρόεδρε έχοντας κατά νου ότι είχα τόσα πολλά στοιχεία να πω, έκανα αξιοσημείωτη προσπάθεια και προσπάθησα να αντικατοπτρίσω εδώ τις ιδέες όλων. Ευχαριστώ. Εσείς ε, μάλλον κάνατε το παγκόσμιο ρεκόρ εδώ στο Κοινοβούλιο. Κανέναν ε, δεν ξέρω που να μίλησε 29 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα συνεχώς. Έτσι λοιπόν, ας ε, περάσουμε τώρα στη συζήτηση με τους διάφορους βουλευτών. Καταρχήν, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερος και όλους τους προσκεκλημένους που συμμετέσχουν στην σημερινή ακρόαση και που έλαβαν το λόγο για να εξηγήσουν τις απόψεις τους για την περιφερειοποίηση, απόψεις που σίγουρα είναι πολύ σημαντικές στα πλαίσια της προσπάθειας μεταρρύθμισης της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τον, ε, ε, απευθύνεται μάλλον στον κύριο Ριόρνταν. Είπε ο κύριος Ριόρνταν ότι στην βάση της περιφερειοποίησης πρέπει να μπουν οι διάφοροι τομείς της αλίας και ιδιαίτερα κύριε Ριόρνταν αναφερθήκατε στην ε, αλεία μικρής κλίμακας. Μπορείτε να ορίσετε αυτή την μικρή κλίμακα αλία. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σα, ποιο είναι ο ορισμό, πώ ορίζεται η αλία μικρή κλίμακα. Και αν δεν μπορείτε να δώσετε ένα συγκεκριμένο ορισμό, μπορείτε να μα πείτε ποια είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμοστούν για να καθοριστεί αυτή η αλία μικρή κλίμακα. Δεύτερη ερώτηση για τον κύριο Σάμποργκ, ο οποίο μίλησε για την αναγκαιότητα της περιφερειοποίησης στα πλαίσια του προβληματισμού για την Βαλτική θάλασσα και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αποθέματα βακαλάου και επέκρινε μάλιστα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κοινή αλληλευτική πολιτική που ισχύει τώρα. Μπορείτε να μας πείτε αγαπητέ κύριε για ποιο λόγο είναι τόσο επικριτική η θέση σας. Και τέλος για τον κύριο Μπαντιόλα. Μιλώ για, τις, για τους ε, γνωμοδοτικούς περιφερειακούς οργανισμούς Πράγματι η παρέμβασή σας ήταν μακροτάτη και πλήρης λεπτομεριών. Μιλήσατε για, εξηγήσατε μάλλον πώς είναι η παρούσα κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να μάθω εάν οι περιφερειακές, οι περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια είναι έτοιμα όσοι στο μέλλον να αναλάβουν την ευθύνη, στο μέλλον να αναλάβουν την ευθύνη της διαμόρφωσης της αλληλευτικής πολιτικής. Είναι έτοιμα τα όργανα αυτά να συμμετάσχουν στην νομοθετική αυτή διαδικασία που σημαίνει βεβαίως ανάληψη και πλήρους της ευθύνης για την εφαρμογή της προτινόμενης πολιτικής. Είναι έτοιμα τα γνωμοδοτικά αυτά συμβούλια να αναλάβουν την πρόκληση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιράντα. Μιράντα, Μιράντα. Gracias, presidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να απευθύνω με τη σειρά μου χαιρετισμό και το καλωσορίσατε σε όλους τους συμμετέχοντες που έλαβαν το λόγο και ε, ανέπτυξαν τα θέματα με εξαντλητικό τρόπο. Στην πολιτική μας ομάδα είχαμε πολύ, πολλές επαφές μαζί σας. Συμφωνούμε με την θέση μεγάλου μέρους των παρεμβάντων που εξήγησαν ότι η, μετα... η, κοινή, η πολιτική που ισχύει σήμερα είναι υπερβολικά συγκεντρωτική και χρειάζεται μια συνδιαχείριση που είναι και ο καλύτερος δείκτης σωστής διαχείρισης. Ο κύριος Τεκολούνια, παλιός καθηγητής μου έχει επιμείνει στο, στο στοιχείο αυτό. Επίσης, είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε βάθος η αποκεντροποίηση της διαχείρισης της μικρής κλίμακας αλίας. Και αυτή η ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Όρι Όρνταν. Υπάρχουν δείκτες όχι μόνο οικονομικοί αλλά και βιολογικοί και κοινωνικοί και ε, απευθύνομαι και στον κύριο Τρουχίγιο με ποια κριτήρια θα γίνει η αποκεντρωμένη προσέγγιση. Τέλος, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να διατεθούν περισσότεροι πόροι. Δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί πολιτική χωρίς πόρους. Δεν μπορεί κανείς να δράσει, να κάνει γνωμοδοτήσεις, να διαβουλεύσεις χωρίς να έχει επαρκείς πόρους. Και γι' αυτό νομίζω ότι η προσέγγιση των ε, περισσότερων παρεμβαινόντων είναι σωστή. Χρειάζεται λοιπόν μια συνολική προσέγγιση περιβαλλοντική, οικολογική, οικονομική, κοινωνικο-οικονομική, γιατί εν τέλει είναι βέβαιο ότι είστε οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι για την διατήρηση του πλούτου αυτού των αλληλευτικών αποθεμάτων. Η κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους ε, προσκεκλημένους του σημερινού απογεύματος που νομίζω ότι η συμμετοχή τους μας ανοίγει νέους δρόμους για το τι μπορεί να σημάνει η αποκέντρωση στο μέλλον. Παρακολούθησα προσεκτικά τις περισσότερες από τις ε, παρεμβάσεις σας. Ε, η γνώμη σας φαίνεται πως είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι απολύτως πιστική. Το Κοινοβούλιο άλλωστε μοιράζεται αυτή τη γνώμη, διότι θεωρούμε ότι εν μέρη αυτό οδηγεί σε μια επανεθνικοποίηση, αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, τα τεχνικά μέτρα που θα αναλάβουν οι χώρες μέλη κλπ. Ξέρω ότι τα πει από αυτά ο κ. Μπαρδιόλα και απέρριψε αυτή την άποψη. Χρειάζεται λοιπόν συνένεση. Αυτό μου φαίνεται λογικό. Δεν θέλουμε μέτρα τα οποία να έχουν διακριτικό χαρακτήρα, να, να, να προβαίνουν σε διακρίσεις κατά ορισμένων ε, ειδών αλίας, κατά ορισμένων στόλων και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια βάση να γνωρίζουμε τι δεν θέλουμε. Όλοι μας το γνωρίζουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά επίσης την διαδικασία, τι μπορεί να μας οδηγήσει σε καλύτερη τυποποίηση, αποκέντρωση, περιφερειοποίηση, όπως θέλετε, πέστε το. Για το συγκεκριμένο αυτό, θα ήθελα τα πράγματα αυτά να μας βρουν σύμφωνους όλους. Αυτά που είπε ο κ. Σομπρίνο, κατανοώ την γνώμη του, κατανοώ την άποψή του και ελπίζω πολύ οι νομικές υπηρεσίες επίσης να την καταλάβουν. Διότι αυτό που έκανε ήταν να μας δώσει μια νομική ανάλυση και νομίζω ότι είναι μια, μια ε, άποψη η οποία θα μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερη περιφερειοποίηση. Βέβαια ότι και εγώ είμαι νόμο μαθής. Και δεν μπορώ να είμαι βέβαια αν αυτά είναι συμβατά με τις συνθήκες. Έχουμε λοιπόν εδώ σκιαγραφίσει μια διαδικασία που ενδεχομένως μπορούμε να ακολουθήσουμε και μπορεί να αποβεί χρήσιμη για την μελλοντική μας εργασία. Και απευθύνομαι εμέσως και στην κυρία Ρόντουστ. Επίσης, οι απόψεις του κυρίου Μπαντιόλα για τα ΡΑΚ και από του κυρίου Σομπρίνο. Νομίζω ότι τα δύο έγγραφα των δύο ανδρών μπορούν να θεωρηθούν αλληλοσυμπληρούμενα. Πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Κομισιόν, ΡΑΚ, τα κόρε πέρα, ας πούμε, όπως τα λέμε, στο επίπεδο του Συμβουλίου που είναι αυτά που εξήγησε ο κύριος Σομπρίνο και όλη αυτή η διαδικασία, η νομοθετική διαδικασία, η συνήθις τακτική νομοθετική διαδικασία με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά εν προκειμένου αυτό που θα ήθελα να κάνω να ζητήσω να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δέχεται τι προτάσει αυτέ. Επίση, θα ήθελα να βολιδοσκοπήσω τι νομικέ μα υπηρεσίε. Τι γνώμη έχουν στο μέλλον, μπορεί να συμφωνήσουν με τι θέσει αυτέ. Να μα πούν ενδεχομένω ότι είναι συμβατέ με τι ε, συνθήκε. Είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που θεσπίζουν οι συνθήκε. Συμφωνώ και με τον κύριο Σοπρίνο και με τον κύριο Μπαντιόλα. για το δικό σας θέμα κύριε Παντιόλα, δεν είμαι βεβαίω ότι κατάλαβα καλά. Η σύνθεση των μελών των ΡΑΚ θα αλλάξει και αυτή. Θα περιληφθούν για παράδειγμα επιστήμονες, θα περάσει το επιστημονικό στοιχείο, θα εισέλθει στα ΡΑΚ. Τέλος πάντων, εγώ πάντως συμφωνώ με τον κύριο Παντιόλα στα όσα είπε, ότι χρειάζεται να είναι υποχρεωτική διαδικασία για τα ΡΑΚ. Και όπως σωστά είπε και στην έκθεση, Χρειάζεται επίσημη αναγνώριση, βεβαίως μέσα στα νομικά πλαίσια, αλλά και, όπως είπα, επίσημη αναγνώριση. Και αν εν τέλει υπάρξει απόκληση από τις προτάσεις των ΡΑΚ, αυτή, εφόσον λέω υπάρχει απόκληση, η απόκληση αυτή θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Τα όσα ακούσαμε ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Πατιόλα και τον κύριο Σομπρίνο, ιδίω αυτού του δύο εμπεριγνώμονε. Νομίζω ότι αυτά που έχουν καταθέσει μπορούν να αποτελέσουν ένα χάρτη πορεία για μα. Θα ήθελα ακόμη να πω, όπω είπα πριν, την θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθώ επίση και τι νομικέ υπηρεσίε, τη δική μα νομική υπηρεσία. Εάν υπάρχουν νομικέ ενστάσει για αυτά που λέμε ή αν είναι πραγματικά στεγανά. Ευχαριστώ κυρία Πατράου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, λυπάμαι γιατί αναγκάστηκα να αποχωρήσω για λίγη ώρα και να απουσιάσω από αυτήν την ε, τόσο σημαντική ακρόαση, δεν μπορούσα να το αποφύγω. Ε, πήγα σε ένα τριμερή διάλογο. Όπως και η συνάδελφο ε, Κάρμεν Φράγκα θέλω να επιμείνω για κάποια ζητήματα. Συμφωνούμε όλοι με την περιφερειοποίηση. Ε, είμαστε όλοι απογοητευμένοι από τις προτάσεις Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δηλαδή μας αναθέτει και πάλι σε εμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ρόλο να βρούμε καλύτερες λύσεις, τις λύσεις που εκείνη δεν κατόρθωσε να βρει και εδώ έχουμε τους ιδανικούς συνομιλητέ που μπορούν να μας ενημερώσουν, να κατατοδέουν και να επιτύχουμε την περιφερειοποίηση. Ε, είμαστε ε, όλοι σύμφωνοι ότι πρέπει να επιδιώξουμε την ε, περιφερειοποίηση και ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της περιφερειοποίησης φυσικά είναι οι προτάσεις που θα κατατεθούν εν ώψη της μεταρρύθμισης κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο από όλα είναι το εξής. Η, ε, τα περιφερειακά χνομοδοτικά ε, συμβούλια πώς αντιλαμβάνονται αυτόν τον νέο ρόλο του στα πλαίσια της ε, μεταρρυθμισμένης και περιφερειοποιημένης κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Ποιες αλλαγές πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν ως προς τη σύνθεσή τους ή τον τρόπο λειτουργία τους. Ε, πώς ε, θα υπομισθούν τις νέες ευθύνε τους. Πώς θα προετοιμαστούν για να αναλάβουν τον νέο τους ρόλο στο πλαίσιο της αναπόφευκτης περιφερειοποίησης. Θα ήθελα επίσης να ακούσω από πλευρά του εκπροσώπου των ε, Περιφερειακών Οχνομοδοτικών Συμβουλίων το εξή. Με ποιο τρόπο ε, θα κατοχυρώσουν την περιφερειοποίηση ή τα γνωμοδοτικά συμβούλια και αναφέρομαι εδώ σε κάποιες επικρίσεις που έχουν ακούστη ότι παρά είναι ανομοιογενή αυτά τα γνωμοδοτικά συμβούλια ε, για να λειτουργήσουν με νέο τρόπο. Ποια κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αποφασίσουμε αν θα είναι σε θέση να λάβουν αυτό το ρόλο ε, τα συμβούλια. Δεν θέλω φυσικά να πολλαπλασιάζονται οι διοικητικές ε, δομές, αλλά σε αυτό το πλαίσιο ίσως θα έπρεπε να επανασχεδιάσουμε την ίδια τη λειτουργία των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων. Ε, τελευταίο θέμα που θέλω να γύρω από τη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά. Συζητούμε ε, πάρα πολύ για την πολυεπίπεδη ε, διαχείριση, multi-level governance. Δεν είναι μια πρόταση των συνθήκων, ειδικά για τον τομέα της αλίας, όπου και μας οδηγεί στην προηγουμένη περίπτωση στην περιφερειοποίηση. Είναι μια γενικότερη πρόταση όπου επιδιώκεται μεγαλύτερη αποκέντρωση, δηλαδή οι εμπλεκόμενοι φορείς σε όλους τους τομείς θα πρέπει να είναι πιο δραστήριοι ε, και να συμμετέχουν ένεργα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς. Στον τομέα της και βάσει του προτύπου της ε, περιφερειοποίησης ε, ποιες δυσκολίες, ε, ποιες ε, προκλήσεις προβλέπετε ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε στο μέλλον και φυσικά στρέφομαι και πάλι στον εκπρόσωπο των περιφερειακών συμβουλίων για την απάντηση. Σας ευχαριστούμε κυρία Πατράου Νέβες. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, οπότε θα ακούσουμε τα μέλη του πάνελ. Επιλέξτε εσείς με ποια σειρά θα παρέμβετε για να απαντήσετε. Ο κύριος Μπαντιόλα θα αρχίσει. Κύριε Μπαντιόλα, μας επιτρέπετε να, μας να δώσουμε τον λόγο στον εκπρόσωπο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Νομικής Υπηρεσίας. Ο Ερνέστο Πένας από πλευράς Επιτροπής ε, θα πάρει πρώτος τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ομολογώ ότι είναι ε, νέα αυτά τα ε, δεδομένα για μένα, όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν έχω ξανακούσει αυτές τις κατηγορίες ότι είμαστε άχρηστοι, ότι δεν κάνουμε τίποτα, δεν είμαστε επιτυχείς ως προς την εκπλήρωση των στόχων που έχουμε θέσει. Τέλος πάντων, Κατά την προετοιμασία ε, των προτάσεων για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτικής αναλύσαμε πάρα πολλά στοιχεία για το ρόλο των ε, περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων. Εξετάσαμε διάφορα πρότυπα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. Ε, η βασική μας μέρη ήταν να μην παραβιάζουμε με τις προτάσεις μας τις διατάξεις της συνθήκης και γι' αυτό χρειάζεται σκέψη. Όλοι πρέπει να προβληματιστούμε ε, και ο ο Σομπρίνο το ανέφερε αυτό. Είχαν κάποιοι την ιδέα να συστήσουν μίνι συμβούλια, μίνι κορεπέρ, ε, άλλες δομές, άλλες ομάδες ε, οι οποίες όμως δεν λύνουν όλα τα προβλήματα διότι δημιουργούν αμέσως αμέσως ε, προβλήματα θεσμικού ε, χαρακτήρα. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποιος θα είναι ο ρόλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα αυτά. Μιλήσαμε για τα μην συμβούλια, μην κορεπέρε με σύνθεση ελάχιστη 10 ατόμων, παραδείγματο χάρη. Πώ ακριβώς θα συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποιο είναι ο ρόλος που θα αναλάβει σε όλα αυτά τα αποκεντρωμένα συστήματα λήψη αποφάσεων. Ίσως ε, θα μπορούσαμε όμως να τα, μας τα ξεκαθαρίσετε λίγο καλύτερα για να μπορέσουμε και εμείς να απαντήσουμε. Δεύτερον, πιστεύω ότι ο καθορισμός συστημάτων ε, λήψης αποφάσεων ε, θα έχει προβλήματα έτσι όπως μας είπε και ο συνάδελφο αν έχουμε ένα είδο μήνυ κορεπέρ, πώ θα διαχειριστούμε τα πελογικά είδη. Αν ε, μου λέει το πελογικό συμβούλιο δεν μπορεί αυτό να περιφερειακοποιηθεί, αυτό θα πρέπει να το δούμε σε συνεργασία με τρίτε χώρε. Ε, εγώ πιστεύω ότι όταν παρουσιάζουμε τέτοια μοντέλα θα πρέπει να ε, συνειδητοποιούμε και περί τίνο πρόκειται. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό όταν ε, μιλάμε για τη δημιουργία ομάδων εργασίας, για τη δημιουργία δομών ε, περιορισμένων ε, σε κάποια κράτη-μέλη κτλ. Στις εντατικέ επαφές που έχει η Κομισιόν με τα κράτη-μέλη υπάρχει ένα θέμα που ανακύπτει συνεχώς, ένας, ένας σημαντικός περιορισμός ε, από την πλευρά πρακτικά όλων των κρατών μελών για να προχωρήσουμε στον τομέα της περιφερειοποίησης και είναι το θέμα της μη αύξησης της διοικητικής πολυπλοκότητας και του διοικητικού άχθου των εθνικών δικήσεων. Το είπε και ο κύριο Βατιόλα, ε, δεν ε, θέλουν νέες πολυπλοκές δομέ, ούτε και εμείς ε, Και τελικά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι την περιφερειοποίηση όλοι τη θέλουμε να την προτείνουμε όχι μόνο για την αποκέντρωση αυτή καθ' αυτή, αλλά και για την απλούστευση. Γιατί η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Βρυξελών είναι κάτι ιδιαίτερο πολύπλοκο και όλοι θέλουμε την απλούστευση. Αν ε, τελικά ε, δημιουργηθούν ε, νέα ε, ενδιάμεσα όργανα που κατά κανένα τρόπο δεν θα καταργήσουν τα σημερινά, δηλαδή όλοι λένε να δημιουργηθούν νέα όργανα, αλλά κανείς δεν ε, είπε ότι θα καταργηθεί η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ε, ή τα ΡΑΚ. Έτσι λοιπόν τελικά τι κάνουμε, απλά προσθέτουμε και άλλα στρώματα διοικητικής περιπλοκότητας. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε εις βάθος πρόεδρε, γιατί η περιφερειοποίηση πρέπει να πλουστεύσει αν ε, τελικά προκύψει αύξηση των άτυπων ή της οργάνων που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, να αναρωτηθεί ίσως κάποιος αν τελικά απλοποιούμε κάτι εδώ. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναφερθούμε στο ρόλο των ΡΑΚ, ε, έτσι όπως ε, περιγράφει από διάφορους ομιλητές υπάρχουν ε, καλές ιδέες που εκφράστηκαν σε σχέση με τα ΡΑΚ. Φυσικά η Κομισιόν προετοιμάζει τώρα ένα έγγραφο το οποίο θα σας το παρουσιάσει και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο αλλά και στα ίδια τα ΡΑΚ για αυτά που είπε ο κύριος Βαντιόλα ως τον ενισχυμένο ε, γνωμοδοτικό ρόλο των ΡΑΚ. Συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι ενισχυμένο ο ρόλος των ΡΑΚ και πρέπει ίσως να το προσέξουμε καλύτερα. Εργαζόμαστε για, επί αυτού και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Παραδείγματο χάρη ιδέα ότι τα ΡΑΚ ε, σχετίζονται με προτεραιότητε, με έρευνα που έχουν μια πιο στρατηγική σχέση με την Κομισιόν. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που μπορούμε να προωθήσουμε. Φαίνονται θετικέ. Προσωπική τοποθέτηση βέβαια. Άλλο θέμα το πώ ε, θα έχουμε διεθνική χρηματοδότηση μέσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Αυτό είναι θέματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ένα σχόλιο Βλέπω στη συζήτηση αυτή και όχι μόνο σε αυτή, αλλά σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε για την περιφερειοποίηση, μια αντίφαση, γιατί αφενός όλοι λένε ότι πρέπει να αποφύγουμε το one size fits all, δηλαδή ότι ένα μέγεθος κάνει σε όλους, δηλαδή ότι Πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική συγκέντρωση, πρέπει να αποφύγουμε να υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο μικροδιαχειριζόμενο που θα εφαρμόζεται αυτόματα σε όλε τι περιφέρειε. Πολύ ωραία, πρέπει να τα αποφύγουμε όλα αυτά. Όταν μιλάμε για τρόπου εφαρμογή για την ε, περιφερειοποίηση, το πρώτο που μα ζητάτε είναι να πούμε με ακρίβεια πώ θα είναι η διαδικασία, ποιο είναι ο ρόλο του κάθε πρωταγωνιστή, ποιο ακριβώ ε, θα αποφασίσει τι. Δεν ε, υπάρχει μια αντίφαση σε όλα αυτά. Δηλαδή θέλουμε να φύγουμε από τη μικροδιαχείριση και το πρώτο που μας ζητάτε είναι να, να μικροδιαχειριστούμε τον τρόπο που θα προσεγγίσουμε αυτή την περιφερειοποίηση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά και τέλος να σας υπενθυμίσω το παράδειγμα του Σκάγκερακ. Αν ε, τώρα η περιφερειοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει να μεταφράζεται σε κάτι απτό και πραγματικό, το παράδειγμα που έχουμε ενώπιόν μας είναι του Σκάγκερακ και ε, προχωρά το θέμα του Σκαγκερέκ, όχι γιατί η Κομισιόν είπε ότι πρέπει να γίνει κάτι και το κατέρτισε η Κομισιόν και έθεσε κάποιου λεπτομερεί κανόνε, αλλά γιατί επειδή οι δύο κρατημέλη και τρίτη χώρα ανέλαβαν την πρωτοβουλία να συμφωνήσουν για ένα νέο σύστημα. Και όταν αυτό γίνεται, η Κομισιόν συμμετέχει και διαδραματίζει το ρόλο τη. Αυτό θεωρώ εγώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην νομική υπηρεσία για να απαντήσει εν συντομία στις ερωτήσεις που ακούστηκαν και κάτι να πω στον πρόσωπο της Κομισιόν. Δεν ήταν γνωμοδο... άποψη της κυρίας Φράγκα αλλά ήταν απόδειξη από όλη την σημερινή συζήτηση. Παρακαλώ, η νομική υπηρεσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω εντάχει να αναπτύξω κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, δίνοντας μια απρόορη απάντηση σε ανησυχίες της κυρίας Φράγκα για το ενδεχόμενο σύσταση αυτών των μήνυ κορεπέρ. Πρώτα απ' όλα, ε, την προσοχή σας στο ότι μας ζητήθηκε από εσά εχθές επίσημη γνωμοδότηση και ακόμη την επεξεργαζόμαστε θα, όσα θα πω λοιπόν ε, είναι υπό την επιφύλαξη της διατύπωσης της, ε, και το περιεχομένου της ε, γνωμοδότησης. Παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η γνωμοδότηση, θεωρώ ότι είμαι ήδη σε θέση να σας πω τα εξής. Από νομικής πλευράς για το θέμα της περιφερειοποίησης πρέπει να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα σε δύο διαστάσεις που δεν αλληλοαποκλείονται αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Πρώτον, υπάρχει μία περιφερειοποίηση ε, όπως αυτή αποτυπώνται στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η νομική βάση σε αυτή την περίπτωση θα είναι το άρθρο 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ασκήσουν κάποιες αρμοδιότητες που υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή όλα τα αλληλευτικά θέματα επανεκχωρεί αν θέλετε αυτή τις αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στα κράτη-μέλη. Αντί να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δρούν τα κράτη-μέλη Άρα οι συνομιλητέ, ε, ή μάλλον ναι, παρόλα αυτά ο συνομιλητή θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι τα κράτη-μέλη. Βάσει τη συνθήκης, ξαναλέω, εκχωρεί η Ευρωπαϊκή της συνθηκη ξαναλεω εκχωρει η ευρωπαικη επιτροπη τις αρμοδιότητές τη. σε άλλους οργανισμού σε άλλες οντότητες λέει η συνθήκη, αλλά εν τέτοιου περιπτώσει ε, τι σημαίνει αυτό, μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν ε, να είναι αυτές οντότητες και δεν ανατίθεται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρμοδιότητες σε οντότητες και οργανισμούς κάτω από το εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι ε, μια πρώτη αρχή. Ε, δεύτερον, Τα κράτη-μέλη ε, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αρμοδιότητες που όπως σας έλεγα ε, συνιστούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ό,τι σχετίζεται δηλαδή με την αλία. Και όπως σας είπα δεν μπορεί η Επιτροπή να συνομιλεί με οντότητες άλλες πέρα από τα κράτη-μέλη. Άρα δεν υπάρχει άλλος νομικός τρόπος, αν θέλετε, παρά να περάσουμε μέσα από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οργανισμοί που δεν είναι κράτη-μέλη για να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειάζεται αυτή η νομική ρύθμιση. Αυτό και μόνο αποκλείει τη δυνατότητα της σύστασης ε, μιας μήνυ κορεπέρ. Θα επανέλθω σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να υφίστανται τέτοιοι οργανισμοί, όμως ε, δεν γίνεται να εξουσιοδοτούνται οι οργανισμοί αυτοί άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι, όπως είπε και ο κύριος ε, Πένας ε, Λάντα, δεν υπάρχει τρόπος να ενσωματωθούν οι μήνυ κορεπέρε όπου ε, συγκεντρώνονται εκπρόσωποι κυβερνήσεων κάποιων παρακτήων κρατών στις θαλάσσιες λεκάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι δίνεται η έγκριση για να ασκηθούν αρμοδιότητες που κανονικά είναι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προ τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή και η δεύτερη πτυχή που ε, ήδη ε, ανέφερα πολλές φορές δεν αποκλεί την πρώτη ε, νομική δυνατότητα, δηλαδή τη δυνατότητα των κρατών μελών να ασκήσουν εξ ονόματο τη Επιτροπή κάποιε αρμοδιότητε, ούτε αποκλεί την ταυτόχρονη ύπαρξη άλλων οντοτήτων που θα μεταφράσουν στην πράξη την περιφερειοποίηση. Όμως θα βασιστούμε ως επιδοπλίστων σε υφιστάμενα πρότυπα διαχείριση των αλλιευμάτων βάσει τη νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, την άμεση αυτή η ανάθεση ε, δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να εφαρμόσουμε το πρότυπο της ε, μικροδιαχείρισης. Όταν ανατίθενται αρμοδιότητες από την Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη για την κατάρτιση, παραδείγματος χάρη πολιετών σχεδίων για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων, όπως εξάλλου προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη, ε, υπολείπονται και κάποιες άλλες αρμοδιότητες που επίσης αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και σε αυτό το πλαίσιο ένα και περισσότερο γίνεται άμεση ανάθεση βάσει μιας ενισχυμένη ε, ε, κανονιστικής ε, δομής όπως το, η ΣΤΕΦΚ, η Τεχνική Επιστημονική και Οικονομική Επιτροπή ΣΤΕΦΚ ή ε, τα CCRs μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, αυτές ε, οι δομές, αλλά ούτως ή άλλως πρόκειται για άμεση ε, άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τους οργανισμούς της. Διότι ξέρετε ότι πέρα από, συνομοθε... πέρα από την νομοθετική της πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνεται βάση των αρμοδιοτητων της ευρωπαικης επιτροπης απο τους οργανισμους της διοτι ξερετε οτι περα απο περα απο την νομοθετικη της πρωτοβουλια η ευρωπαικη επιτροπη δινεται βαση των συνθηκων να ασκήσει αυτό το ρόλο θα ήθελα να προσθέσω μία λεπτομέρεια. Όπως έχουν τώρα τα πράγματα, ο βασικός ε, ε, κανονισμός Υπάρχουν οι διατάξει ε, του άρθρου 4, εδάφιο 2 και επίσης άρθρο 33, όπου ρητά, Υποχρεώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέγει ε, τις νομοδοτήσεις των ε, Περιφερειακών Νομοδοτικών Συμβουλίων καθώς ε, και της Τεχνικής, Οικονομικής και Επιστημονικής Επιτροπής και να τις λάβει υπόψη κατά την προετοιμασία των μέτρων που θα προτείνει. Παραδόξως στην... δεν υπάρχει πλέον αυτή η ρητή διατύπωση στον ε, ε, ισχύοντα βασικό κανονισμό, αλλά δεν βλέπω κανένα νομικό κόλμα γιατί να μην ε, συμπεριλάβουμε και πάλι αυτήν την διατύπωση στο νέο βασικό κανονισμό. Ως προς την εκχώρηση από πλευράς της Επιτροπής Αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη πέρα από αυτά που αναφέρει ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και με στόχο την ενίσχυση των ε, δομών λήψης αποφάσεων Θα κλείσω, Πρόεδρε, συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά θέλω να ολοκληρώσω αυτό το σημείο. Λοιπόν, έλεγα ότι πρέπει να γίνει η διάκριση ανάμεσα στην περιφερειοποίηση, δηλαδή όταν παίρνουν ε, την εξουσιοδότηση στα κράτη-μέλη να δράσουν εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε επίπεδο κρατών μελών ε, σταματάει αυτό. Δεν μπορούμε να περάσουμε σε ένα κατώτερο επίπεδο, σε κάποιον οργανισμό που ανήκει στο κράτο μέλο. Ε, αυτή είναι η μία εναλλακτική λύση και η άλλη εναλλακτική λύση είναι ε, να εμπλακούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί. η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή, τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και, αυτές, και αυτοί οι οργανισμοί θα έχουν μεγαλύτερο ειδικό βάρο στι υφιστάμενε δομέ ε, ε, λήψης αποφάσεων. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε το λόγο στου ομιλητέ για να απαντήσει, ο καθένα να δώσει συγκεκριμένε απαντήσει. Προσπαθήστε παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Sí, acabo de decir. Eh, empezamos, ya digo, intentando ser muy sintético. Λοιπόν, ε, παρακαλώ προσπαθήστε να είστε πολύ συνθετικοί. Στις απαντήσεις ο κύριος Μπαριόλη καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ στα πέντε μου λεπτά και έχοντας κατά νου ότι είναι εδώ και ο κύριος Ράινερ από το ΡΑΚ της Βαλτικής και ο κύριος Μπαρτιάστρων από το Βορειοανατολικό ΡΑΚ. Εγώ θα ήθελα να δώσω και σε αυτούς ε, το λόγο, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να συμμετέχουν στη συζήτηση. Μάλιστα, βεβαίως. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν ε, θα ήθελα σε καμία περίπτωση να σχολιάσω αυτή την έξοχη παρουσίαση του κυρίου Μπαντιόλα, ε, διότι ε, πραγματικά πηχούνται οι απόψεις όλων των γνωμοδοτικών συμβουλίων. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια επιμέρους ζητήματα. Δεν θα σχολιάσω την τροποποίηση των συνθήκων. Είναι πολύ περίπλοκα αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα μόνο να μιλήσω ε, για την ε, διάσταση της ε, επανεθνικοποίησης που είναι ένας εκείνος που λογεύει με αυτές τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι στιγμή η ελευτική πολιτική είναι αντικείμενο διαχείρισης του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς θέλουμε να δοκιμάσουμε όμως μία νέα πολιτική και όταν ακούμε την περιγραφή της διαδικασίας ε, τη ε, πρακτική που πρέπει να αναπτυχθεί για να μπορέσουν να ληφθούν ε, αποφάσει με ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων μα φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και νομικά δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε, υπάρχουν διαφορετικά τοπικά πρότυπα. Εγώ πιστεύω σε αυτό και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν ανυπέρβλητα εμπόδια για την επικοινωνία αυτών των οργάνων. Όμω υπάρχει μία έλλειψη ακόμη και αν ε, υποβάλλουμε ένα τέτοιο σχέδιο συνεργασίας ε, των ε, περιφερειακών ε, συμβουλίων και ενισχύσουμε δηλαδή τη δομή της μικροδιαχείρισης μπορεί να γίνουμε πολύ αντιπαραγωγικοί όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι και αυτό θα έχει σημαντικότατες επιπτώσεις για τα πολυετή προγράμματα διαχείρισης. Ε, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη ε, κατά το δοκούν. Όμως πρόκειται για μια σημαντικότατη ε, έλλειψη στην όλη διαδικασία. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η νέα πρόταση συνεπάγει το μεγαλύτερο γραφειοκρατικό άχθος ε, και σπέβδουν να πούν ότι δεν χρειαζόμαστε περιφερειοποίηση και ακυρώνεται παραδείγματος χάρη το Balt Fish. Μα είναι πολύ καλή πρωτοβουλία, αλλά ούτως ή άλλως υπάλληλοι είναι από χώρες ε, ε, που περιβάλλουν τη Βαλτική και σίγουρα δεν είναι ε, οι επαγγελματίες του κλάδου. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ένα φόρουμ όπου μπορούμε πραγματικά να συζητήσουμε τα θέματα μικροδιαχείρισης. Τουλάχιστον υπάρχει ένα βήμα όπου κανείς δεν μπορεί να εκθέσει πλήρως την άποψή του. Πήρατε το παράδειγμα του Σκάγκερακ ε, και να, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου υποχρεώνονται ε, οι ε, διαχειριστές να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές για τις απορρίψεις, παραδείγματος χάρη. Η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φινλανδία υποχρεώθηκαν λοιπόν χωρίς καν ακουστεί η φωνή της βιομηχανίας να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο και αυτό συμβαίνει και σε πολλά άλλα περιφερειακά σύμβουλια Γι' αυτό χρειαζόμαστε την ε, περιφερειοποίηση. Πάντως, ε, κλείνοντας θα σας πω ότι για να βοηθήσουμε ε, την κατάσταση, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, αλλά, και, αλλά τα κράτη-μέλη που πρέπει να δραστηριοποιηθούν κατά αυτήν την προπαρασκευαστική περίοδο για να περιγράψουμε την πρακτική που επιθυμούμε να εφαρμοστεί διακόπτει ο Πρόεδρος ε, τον ομιλητή. Παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομος. Κύριε Πρόεδρε, ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Απλώς θα υποστηρίξω τα όσα μόλις είπε ο συναδελφός μου. Το κυριότερο είναι η governance, η διακυβέρνηση. Πρέπει να δούμε ποιο επίπεδο αυτή της διακυβέρνηση μπορούν, ε, ε, μπορεί να στηρίξει τα ΡΑΚ. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε προσεκτικά πώς θα λαμβάνονται υπόψη οι γνωμοδοτικές αυτές συμβουλές και βέβαια τα ΡΑΚ θα χρειάζονται να έχουν στη διάθεσή τους και κάποια μέσα ώστε οι γνωμοδοτήσεις αυτές να καθίστανται δεσμευτικές. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να προσφέρουμε κάποιες συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και αυτές μπορούν να ληφθούν υπόψη ή όχι. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ώστε να κινηθούν προς την κατεύθυνση να γίνουν δεσμευτικές οι γνωμοδοτήσεις αυτές, τουλάχιστον. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τη σειρά. Αν συμφωνείτε, ο κύριος Σόρι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε όντως για ορισμούς, νομίζω ότι η συζήτηση θα γίνει μακρότατη, ακαδημαϊκή και άνευ αποτελέσματος. Σε όλη την Ευρώπη θα δούμε ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί και όροι. Στα αγγλικά small scale, οι Γάλλοι λένε πέσο artisanal, δηλαδή βιοτεχνική αλία, επίσης μικρή αλία, οι Ισπανοί λένε πέσκα χώρα και όλα αυτά είναι όροι που ταιριάζουν στο τοπικό πλαίσιο. Ενώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι μας χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Μας ενδιαφέρει η αλληλεία μικρής κλίμακας διότι θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής μας και δεύτερο χρειάζονται οπωσδήποτε διαχείριση οι αυτέ. αυτές. Άρα χρειαζόμαστε έναν ορισμό που να μας επιτρέψει να καθορίσουμε για ποιο πράγμα μιλούμε για λογαριασμό των, των στόχων μας πολιτικής και πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τον συγκεκριμένο ε, τομέα. Ποιοι είναι οι, στόχοι της πολιτικής μας. Θέλουμε λιγότερη επιρροή στο περιβάλλον, χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων, οι, μικρές, οι μικρής κλίμακας αλίας έχουν οικονομική σημασία για τις τοπικές κοινότητες και θα χαθούν πολλά εάν χαθούν αυτές οι αλληλίες μικρής κλίμακας. Αναγνωρίζουμε ότι οι αλληλίες μικρή κλίμακα είναι ανθεκτικές και προσφέρουν ανθεκτικότητα στι τοπικές κοινωνίε, διότι έχουν γνώση και αποτελούν τρόπου ζωής που αξίζει να τους υπερασπιστεί κανεί. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι έχουν και τρόπους αυτοδιαχείρισης οι αλληλίες μικρά κλίμακα που μέχρι τώρα αποδείχτηκαν εν το χρόνο επιτυχημένες και μάλιστα και εν ώψη του ανταγωνισμού άλλων χρηστών των ίδιων πόρων, δηλαδή των ε, ενδεχομένω των ε, ε, αλλιών μεγάλη κλίμακα ή θαλάσσιων αιωλικών πάρκων κλπ. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που πρέπει να αναζητήσουμε είναι μια προσέγγιση πλαισίου. Να καθορίσουμε δηλαδή τις αλλιές μικράς κλίμακας που να μας επιτρέψει να καθορίσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία να μπορούν να εφαρμόζονται στο τοπικό ή στο περιφερειακό επίπεδο. Διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2009 μια συνάντηση στις Βρυξέλλες με συμμετοχή εκπροσώπων κοινοτήτων μικρής κλίμακας αλλιών από 7 ή 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και στο ανακοινοθέν που εξέδωσαν είπαν ότι ο ορισμός των αλλιών μικρής πρέπει να γίνει στο πιο κατάλληλο επίπεδο, είτε αυτό είναι περιφερειακό, εθνικό ή τοπικό. Αυτοί οι ορισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τη γεωμορφολογία. Επίσης τεχνικές πτυχές όπως την αλληλευτική ικανότητα, περιβαλλοντικές επιλεξιμότητα, χαμηλές απορρίψεις, χαμηλές δηλαδή σε ποσότητες απορρίψεις και ούτω καθεξής. Επίσης κοινωνικά θέματα, αξιοπρεπή εργασία, ε, σημαντικά μερίσματα, δηλαδή απόδοση κερδών και επίσης τα θέματα κυριότητας. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε λοιπόν να εξετάσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε τρία ή τέσσερα σύνολα χαρακτηριστικών, τα οποία θα αναφέρονται στην διαρθρωτική φύση, στο μέγεθος, μήκος, τονάζ υποδύναμη η κιλοβάτ του σκάφους και το είδος των αλευτικών εργαλείων που χρησιμοποιεί. Επίσης, το βελινεκές, το δηλαδή πόσο μέχρι που μπορεί να φτάσει το σκάφος, καθώς και τον τόπο που έχει την έδρα του, την απόσταση από την ακτή, το χρόνο που μπορεί να περάσει στη θάλασσα. Επίσης, έναν αριθμό κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων που να μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την κοινωνική σημασία της δραστηριότητας αυτής. Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το είδος κοινοτήτων όπου έχει τη βάση του το σκάφος, το μέγεθος της επιχείρησης, την κυριότητα της επιχείρησης, αν είναι οικογενειακή, αν είναι συνεταιριστική, αν είναι κάποια κοινοπραξία και ούτω καθεξής. Και μετά μπορούμε να εξετάσουμε και άλλα κριτήρια που μπορούν να εφαρμοστούν και να μας επιτρέψουν να εξετάσουμε τις αλλίες αυτές με καλύτερο τρόπο, δηλαδή την εποχιακή διαφοροποίηση των ε, αλλιευτικών εργαλείων, τις παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης της αλλίας, δηλαδή κλειστές εποχές, κλειστές περιοχές, άνοιγμα σε διάφορα είδη, σε διάφορες εποχές του χρόνου και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την προσέγγιση πλαισίου και ο ρόλος της Κομισιόν θα πρέπει να είναι να δώσει τα κριτήρια και τις αρχές που θα πρέπει μετά να εφαρμοστούν στο τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η δεμία, αν θέλετε να μιλήσουμε για ορισμούς, θα καθίσουμε εδώ τρεις-τέσσερις ώρες ακόμη. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα θα πάρει ο κ. Στρουχίγιο και να προσπαθήσουμε να περιοριστούμε γιατί αφαιρούμε χρόνο από τους επόμενους ομιλητές. Και πάλι Πρόεδρε ευχαριστώ. Θα σεβαστώ το χρόνο γιατί υπάρχουν ε, και κάποιοι ομιλητές ε, που πάνω κάτω είπαν αυτά που έθεσα και εγώ, κάπω καλύφθηκα. Εμείς, ε, αν μιλήσουμε για περιφερειοποίηση, ακολουθήσαμε τον ορισμό της λέξης, αλλά κατανοούμε ότι η κοινή ελευτική πολιτική, όπως ορίζεται, είναι κοινή για όλους. Και στα πλαίσια αυτού του εύρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολλές αποχρώσεις πρέπει να αποκεντρωθεί η λήψη αποφάσεων και να, καθιστού, να κατασταθούν υπεύθυνοι οι πρωταγωνιστές ε, σε πρώτο πρόσωπο και μιλώ για τη διαχείριση, για το περιβάλλον, για την οικονομική βιωσιμότητα, την κοινωνική βιωσιμότητα, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές. Και σε ό,τι αφορά στο ρόλο που πρέπει να έχουν ε, τα ΡΑΚ, όπως εξήξα προηγουμένως, νομίζω ότι είναι θετικά και πρέπει να ενισχυθούν αλλά πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και κυρίως πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση. Πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους για να μπορούν να λειτουργούν. Γιατί αυτή είναι η βούληση και όσον παίρνουν στον ΡΑΕ, καλά πρέπει να δούμε και ποια δυνατότητα θα δοθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, από τα ευρωπαϊκά όργανα, έτσι ώστε να μπορέσουν τα ΡΑΚ να είσαι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Επίσης κατανοούμε ότι οι κοινωνικοί παράγοντες είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μιλώ, για την υπεραστηνική κοινότητα, για τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, γιατί να μιλάμε για αποκέντρωση σημαίνει ότι θα μιλήσουμε για όλη την κοινή ελευτική πολιτική και για τους παράγοντες, για τους πρωταγωνιστές που την επηρεάζουν. Δηλαδή είναι σαν να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα και θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι συνομιλητές. Δεν θα μας φαινόταν ιδιαίτερα σκόπιμο να μειωθούν ε, υπερβολικά τα περιφερειακά, συγγνώμη, τα γνωμοδοτικά όργανα. Αλλά ε, θα πρέπει να ενισχυθούν με τα κατάλληλα μέσα. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομικό ρόλο εμείς ε, δεν θέλουμε να έχουν ε, έναν ε, οργανικό ρόλο, αλλά θέλουμε το όργανο αυτά να είναι γνωμοδοτικά. Όμως οι γνωμοδοτήσεις τους να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Δηλαδή, φυσικά δεν μιλάμε για νομοθετικά κείμενα, αλλά θέλουμε να είναι δεσμευτικές οι γνωμοδοτήσεις αυτές και να καθορίζουν την ε, λήψη αποφάσεων ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τρουχίγιο, τον κύριο Σομπρίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως εγώ να μην ε, τα μπόρεσα να τα εξηγήσω όλα στα 10 λεπτά που είχα για να προσπαθήσω να ορίσω τι είναι αυτές οι επιτροπές που πρότεινα στην παρεμβασή μου για την ε, περιφερειακή διαχείριση της Αλίας. Και γι' αυτό αποκλίνω από αυτό που σκέφτεται η Κομισιόν και επίσης ε, δεν συμφωνώ ακριβώς με όσο επινομική υπηρεσία. Εγώ πρότεινα ένα μηχανισμό απλούστευσης να εισαγάγουμε, όχι ένα καινούριο όργανο στη διαδικασία υιοθέτηση τη λήψη αποφάσεων. Γιατί όταν ε, είπα τι είναι αυτή η περιφερειακή ε, Νομοδοτική Επιτροπή δεν θεωρούσα ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, αλλά πρέπει να περιορίσουμε αυτούς που διαφε... σε αυτού... η συμμετοχή να περιοριστεί σε αυτούς που ενδιαφέρονται άμεσα για ένα είδος ε, αλίας και σε μια συγκεκριμένη λεκάνη θαλάσσια. Για... Αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί ο τρίτος τίτλος του τρίτου τμήματο τη πρώτη κομισιόν δεν λέει τίποτα. Είναι άδειο. Μόνο περιφερειοποίηση λέει. Και πώ άκουσα εγώ εδώ, κανένα δεν έδινε τον ίδιο ορισμό στην περιφερειοποίηση. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε για περιφερειοποίηση, ας δώσουμε περιεχόμενο σε αυτό. Τουλάχιστον, ας δώσουμε έναν ορισμό. Πού καλύτερα να το πράξουμε αυτό από ότι στο άρθρο 5 στην πρώτη κανονισμού για να λέμε ότι ε, την περιφερειοποίηση τη ε, πολιτικ της πολιτικής εννοούμε τα εξή. Και έτσι θα γνωρίζουμε σε ποια ώρα κινούμαστε. Γιατί αν κατάλαβα καλά τον εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας ε, της Κομισιόν δεν μιλούσε για περιφερειοποίηση. Μιλούσε για γεωγραφική αποκέντρωση όταν ε, έλεγε ότι δυνάμει το Άρθρο 2 δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα από τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα από τα κράτη-μέλη. Απλώς λέω ότι πρέπει να απασχοληθούν με αυτό το θέμα αυτά τα κράτη-μέλη που τα ενδιαφέρει το θέμα πάρα πολύ επειδή θα βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη λεκάνη ή επειδή θα ασχολούνται με τη συγκεκριμένη αλία. Όχι δηλαδή να συμμετέχουν κάποιοι για κάτι που δεν θα τους ενδιαφέρει. Αυτή είναι η απόψή μου. Και σε ό,τι αφορά τώρα τη σύσταση αυτή τη μήνυ κορεπέρα ή τη σύσταση των ομάδων εργασία, αυτό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχουν 200 σώματα τη εργασία. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει και μια ομάδα εργασία για την περιφερειακή διαχείριση τη Ελία. Και σε ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα εξαλείψουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου θα συνεχίσει να είναι όσο έχει. Βρισκόμαστε στα πλαίσια της τακτικής ε, νομικής διαδικασίας και θα δρούσε όταν το αναλογεί, δηλαδή τη στιγμή που φτάνει η πρωτοβουλία της Κομισιόν. Αν βρισκόμαστε έναντι μια ειδική διαδικασία, τότε θα είναι ειδική διαδικασία και το Κοινοβούλιο έχει το ρόλο που έχει. Και που όλοι γνωρίζουμε. Και σε σχέση με τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα καθιστούσε πιο αποτελεσματικά τα ΡΑΚ, γιατί ε, πριν να συμμετέχει η Επιτροπή η γνωμοδοτική στη διαδικασία και λέω συμμετέχει όχι να λάβει την τελική απόφαση, η τελική απόφαση θα τη λάμβανε το ίδιο το Συμβούλιο. Δηλαδή στη συμμετοχή θα έπρεπε να ακούσει, θα έπρεπε να λάβει υπόψη την ε, προκαταρκτική γνωμοδότηση του ΡΑΚ, του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, που θα μπορούσε μάλιστα και να ε, πάει ακόμη πιο πέρα μέσα από αυτή την επίσημη αναγνώριση που αναφέρεται. Έτσι λοιπόν, Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι επιτροπές ε, θα μπορούσαν ε, να είναι μία οδός προς διερεύνηση για να μπορέσουμε να δώσουμε συγκεκριμένο νόημα και περιεχόμενο στην περιφερειοποίηση. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ρόντου, τηλεοπρόεδρος, για να κλείσουμε αυτό το πρώτο πάνελ. Στην ουσία θέλω μόνο να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Πράγματι ακούστηκαν πολλές καλές ιδέες, έχω σημειώσει πολλές θα τις εξετάσω προσεκτικά. Βεβαίω επίσης τα έγγραφα που υπέβαλαν οι διάφοροι προσκεκλημένοι μας και θα δω ποια από αυτά μπορούν να περιληφθούν στον βασικό κανονισμό. Συμφωνώ μαζί σας ότι όλοι θέλουμε περισσότερη περιφερειοποίηση. Θεωρώ επίσης ότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε υπεύθυνη στοχοθέτηση για ό,τι αφορά την περιφερειοποίηση. Νομίζω συμφωνούμε επίσης ότι πρέπει να πιστούν οι χώρες μέλη να εφαρμόσουν τους στόχους. Σημαντικό μου φαίνεται και το εξής. Μπορεί κανείς να κρίνει, να επικρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο θέλει, αλλά αν θυμούμε καλά, στην αρχική σκέψη της Κομισιόν είχε ακουστεί ότι και η ίδια η Επιτροπή ήθελε πολύ περισσότερη περιφερειοποίηση από αυτήν που τελικά κατέληξε να περιλάβει τις προτάσεις της και αυτό βέβαια έχει σχέση με το γεγονός ότι η δική της νομική υπηρεσία έχει διαφορετική γνώμη. Δεν μπορείτε να αναμένετε να αντιταχθούμε στις νομικές μας υπηρεσίες και γι' αυτό είμαι πολύ ικανοποιημένη που το Κοινοβούλιο ανέθεσε στη δική μας πάλι νομική υπηρεσία να κάνει τη σχετική μελέτη. Και εκεί ίσως αποδειχθεί ότι έχει πάλι διαφορετική άποψη. Αυτή την άποψη θα πρέπει να την εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και νομίζω ότι στο τέλος πια της προσπάθειάς μας θα προκύψει μια πολύ λογική ε, δομή. Είπα και στην αρχική μου εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι θεωρώ ότι τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια πρέπει να συνδεθούν με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να αποδώσουν. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε όντως ένα ακόμα επίπεδο αρμοδιότητας, δηλαδή μια επιτρεπή, περιφερειοποίησης. Ίσως όλα αυτά μπορούν να λυθούν στο επίπεδο των ΡΑΚ. Και εν τέλει νομίζω πάντως ότι στους γενικούς στόχους συμφωνούμε όλοι. Ευχαριστώ κύριε Ρόντουστ. Ευχαριστούμε κύριε Ρόντουστ. Λοιπόν, να περάσουμε χωρίς χρονοκριβή στο δεύτερο πάνελ που φέρει τον τίτλο Η Στόχη και τα εργαλεία μιας περιφερειοποιημένης σκάλπα». Θα έχουμε δύο παρεμβάσεις εδώ, καταρχήν από τον κύριο Μέκλ Κίτινγκ και δεύτερη από τον ε, κύριο Κράν που βρίσκονται Oh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και τα μέλη της Επιτροπής που μου δίνουν την ευκαιρία ε, να σας μιλήσω σήμερα. Ε, είμαι εκτελεστικός διευθυντής ε, του PAEM, που είναι το Συμβούλιο Ελίας στο Δουβλίνο. Εδώ και 60 χρόνια ασχολούμαστε με την ανάπτυξη του κλάδου στην Ιρλανδία και έχουμε μακρά εμπειρία, λοιπόν. Επίσης, έχω ε, ε, διατελέσει σύμβουλος για την προηγούμενη μεταρρύθμιση το 2002. Επίσης, έχω υπηρετήσει 7 χρόνια στην Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή της ΤΕΦΚ. Μεταξύ άλλων, καλούμαστε εδώ να εξετάσουμε τους στόχους της νέας πολιτικής περιφερειοποίησης ε, της αλληλευτικής πολιτικής και μου κάνει εντύπωση που άκουσα τόσες πολλές επικρίσεις στο πρώτο πάνελ. Αν δεν έχετε αποφασίσει με ποιο τρόπο θα το κάνετε, δεν θα ξέρετε ποια μέτρα να συμπεριλάβετε, ε, δεν θα ξέρετε πώ ακριβώ πρέπει να γίνει. Όλα αυτά συναποτελούν το πακέτο. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την συζήτηση και άρα θα προσαρμόσω και τα δικά μου σχόλια αναλόγω. Ποια είναι η ουσία έχουμε μία δέσμη πραγμάτων που θα μπορούσαμε ενδεχομένω να συμπεριλάβουμε στη νέα περιφερειοποιημένη αλληλευτική πολιτική πολιετή, διαχειριστικά προγράμματα παραδείγματο χάρη. Από μόνο του αυτό είναι ένα περίπλοκο θέμα, αλλά σίγουρα ε, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια συμμετέχουν σε αυτό. Επίση, έχουμε την χορήγηση πρόσβαση ε, ε, στι ζώνε αλληλεία, τεχνικά μέτρα και το ρόλο τη ίδια τη Ε, θα ήθελα να αρχίσω από αυτό. Δυστυχώ δεν αναφέρεται στο νέο σχέδιο του βασικού κανονισμού και αυτό είναι λάθο κατά τη γνώμη μου. Ορισμένοι μπορεί να θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε γιατί είναι τόσο ενσωματωμένη στη διαδικασία που δεν πρόκειται να ακυρωθεί ο ρόλο τη. Εμπιστευτείτε μου, θα πρέπει για να διατηρηθεί ο ρόλο τη να αναφέρεται ρητά η Επιστημονική, ε, Τεχνική και Κοινωνική Επιτροπή. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Ε, νομίζω ότι ξέρουμε όλοι τα βασικά στοιχεία της συζήτηση. Ε, τώρα καλύπτουμε μια θαλάσσια περιοχή που εκτίθεται από τη Μεσόγειο μέχρι τη Βαλτική ή και παραπάνω, πιο βόρεια. Ε, το στοιχείο κλειδί της συζήτηση είναι ότι υπάρχουν κάποια αυτονόητα πράγματα. Είτε μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, είτε για τα δυτικά της Σκοτίας, είτε για τη Μαδέρα, όπως το MSY, η οικοσυστημική προσέγγιση και ούτω καθεξής. Αυτές είναι αυτοί είναι σταθεροί συντελεστέ, ε, δεν αλλάζουν και το ερώτημα που πρέπει να μα απασχολήσει για την περιφερειοποίηση είναι ποιο είναι ο πιο αρμόδιος ε, για να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες. Πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό. Ε, επίσης, είναι τόσο μεγάλη η περιοχή που δεν μπορούμε μέσα από ένα μόνο εργαλείο να ρυθμίσουμε τα προβλήματα. Ε, ας πάρουμε το ψαρά στην Ελλάδα και αν το συγκρίνουμε με το ψαρά στη Γαλλία θα συνειδητοποιήσετε πόσες ε, διαφορές ε, υπάρχουν. Υπάρχουν διαφορές και στην νομοθεσία. Βλέπετε εδώ από το Eurlex ε, την τεκμηρίωση, αλλά πάντως θα πρέπει να έχουν τα μέσα ε, αυτοί που καλούνται να κάνουν την μικροδιαχείριση θα πρέπει να έχουν και τα πετούμενα μέσα στη διάθεσή τους. Υπάρχουν βασικά ζωτικά σημεία, επ' αυτών συμφωνούν όλοι, αλλά άλλο πράγμα είναι τεχνικές λεπτομέρειες και πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσετε για αυτά. Αλλά θα πρέπει να αναρωτηθείτε, υπάρχει καλύτερος τρόπος για να διαχειριζόμαστε ελιεύματα σε σχέση με σήμερα δηλαδή. Πάντω ε, πρέπει να έχουν διδακτορικό στην νομική όποιοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο να καταλάβουν όλα, όλα αυτά τα νομοθετήματα. Δηλαδή με ξεπερνάει το πώς συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσει. Εγώ ίδιο δεν τα καταφέρνω να τα παρακολουθήσω. We are top down, we are centralized and we είναι, ε, κάνουμε την μικροδιαχείριση, είναι κεντρικό το σύστημα, αλλά δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κληρονόμησε το σύστημα, παρά είναι υπερβολικό, ε, αυξάνεται καθημερινά ο όγκος της νομοθεσίας και αυτή η υπέροχη ιδέα ότι θα έχω, ε, ότι είναι απλώς αυτός ο βασικό κανονισμός 850, μα τι λέμε, Εάν θέλετε να πάτε να ψαρέψετε στην ε, θάλασσα δίπλα στην Ιρλανδία, έχουμε τα τεχνικά μέτρα, τα ειδικά μέτρα για τον μπακαλιάρο. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμορφωθεί κανείς. Ε, δεν ισχυρίζομαι ότι ισχύει αυτό, αλλά υπάρχουν ισχυρισμοί ότι και οι ψαράδες θα σας το πούν ότι με, αυτήν την, ε, με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές που τους δίνετε ε, χάνουν την εμπιστοσύνη που έχουν σε εσά ε, και όπου και να πάτε όλοι θα σας πούνε ότι δεν ισχύουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμοί. Αυτή είναι η κατηγορία. Δεν λέω ότι ευσταθεί, αλλά έτσι αντιλαμβάνεται ο κλάδος το θέμα παρά είναι κεντρικό το σύστημα, παρά είναι περίπλοκο και δεν ακούγεται η φωνή τους. Το Περιφερειακό Νομοδοτικό Συμβουλίο είναι ο μοναδικός οργανισμός όπου μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους. Ας δούμε τώρα την αναθεώρηση το 2002 τη κοινή αλληλευτική Πολιτική και α αναρωτηθούμε ποια ήταν η προσθέμενη αξία τη. Δεν χρειάζεται να είμαστε υπερβολικά επικριτικοί. Τώρα μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η μεταρρύθμιση του 2002 έριξε τους σπόρους τώρα οι οποίοι αρχίζουν να καρποφορούν σε διάφορου τομεί ε, πάντως, ε, ε, ε, κάποιοι ε, ριζοσπαστικοί παράγοντες αντιτάχθηκαν σε αυτή την απλή ιδέα ότι δηλαδή αντί να καθόμαστε να κοιτιόμαστε θα κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι μαζί με τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις για να αποφασίσουμε. Τότε ήταν, δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η ιδέα, ε, θεωρείται ανατρεπτική και τώρα 8 χρόνια, 9 χρόνια μετά ε, συνειδητοποιούμε ότι μπορούμε να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή. Όλα τα κράτη μπορούν να συνεργαστούν αρκεί να έχουν έχουν το πλαίσιο. Έχετε αυτή ή την άλλη επιλογή. Ε, μπορεί να είναι και οι δύο δυσάρεστε επιλογέ, αλλά αυτή είναι η επιλογή και οι, ε, τα ΡΑΚ μπορούν να πάρουν σωστέ ε, αποφάσει. Πώ λοιπόν μπορούμε, μπορούν να αποδώσουν οι προσπάθειέ μα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο τελευταίο ομιλητή, ότι όλα αυτά ε, τα νομικήστικα μα ξεπερνούν. Αυτό που δεν θέλουμε είναι η ε, επανεθνικοποίηση. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το σχόλιο, διότι όταν. Ε, ένα λεπτάκι γιατί πάτησα λάθος κουμπί. Όταν λοιπόν αρχίζουμε να ζητούμε αυτό το θέμα, συνειδητοποιούμε ότι ε, αναπόφευκτα θα εξετάσουμε και το βασικό κανονισμό. Σήμερα ε, έγινε μια ευρύτατη συζήτηση. Εγώ θέλω να την ε, επανεστιάσω σε αυτά που έχουμε μέσα στο κείμενο. Υπάρχουν τρει ε, τίτλοι, τρία κεφάλαια. Ένα τα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεύτερον περιφερειοποίηση και τρίτον εθνικά μέτρα. Δεν θα ασχοληθώ με τα εθνικά μέτρα διότι σχετίζονται μόνο με τα σκάφη που φέρουν την σημαία του κράτους ε, ε, αλλά τέλος πάντων δεν έχει αυτό σημασία. Θα περάσω τώρα στην περιφερειοποίηση, στο σχετικό κεφάλαιο. Αυτό έχει σημασία. Αναφερθήκατε εσείς στο άρθρο 2 της Συνθήκης, ε, Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεξής. Λοιπόν, ε, όταν πάτε σε αυτό το κεφάλαιο βλέπετε δύο πράγματα. Πρώτον, ποιοι είναι οι στόχοι της περιφερειοποίησης, μα αναφέρονται πολιετή προγράμματα και τεχνικά μέτρα. Συμφωνώ. Αλλά ο διάβολο κρύβεται πάντοτε στι λεπτομέρειε. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και συνειδητοποιήστε ότι δεν πρόκειται για περιφερειοποίηση, πρόκειται όντω για επανεθνικοποίηση, διότι όπω ακούσαμε, ο μοναδικό οργανισμό ε, είναι ε, τώρα και κατεβαίνουμε λίγο παρακάτω στο άρθρο 2 και βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι ε, ε, τα μόνα εξουσιοδοτημένα για να πάρουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν την εθνική νομοθεσία και θα εφαρμόσουν ε, στη συνέχεια. ακολουθεί μια διευκρίνηση και θα επανέλθω σε αυτή. Αλλά πάντως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή η ερώτηση που κάνετε δεν σας δίνω απάντηση. Αν πρόκειται όντως για περιφερειοποίηση ή είναι επανεθνικοποίηση. Δρούν τα κράτη-μέλη μεμονωμένα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή πρέπει να συνοηθούν με τους υπόλοιπους ε, με τους οποίους μοιράζονται και τα αλλιεύματα. Ε, ποιος ακριβώς, με ποιον ε, μιλάμε. Δεν αναφέρεται, ε, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα οι συνομιλητές και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται το διάλογο. Σας δούμε κάπως τους στόχους. Αν δείτε τώρα τα δύο άρθρα αυτού του κεφαλαίου, το ένα σχετίζεται με τον πολιετή σχεδιασμό και εδώ ε, ρυθμίζουμε πολύ λεπτά ζητήματα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όντω, ε, οικοσυστημική προσέγγιση, οι δείκτε, ε, τα τεχνικά μέτρα, οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αλλά όταν μιλάμε για την επιλογή των ειδών του εξοπλισμού, για τα τεχνικά μέτρα, όλα αυτά ωραία και τέλεια είναι, αλλά δεν αρκούν. Α πάρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θα σα πει ο ψαρά ε, ότι έχετε ε, στην Ιρλανδία για τα μικρότερα, μικρότερο μέγεθο ματιού δικτυού, γιατί χρειάζεται αυτό για τα είδη που αλλιεύονται εκεί. Τι εννοώ. εννοώ ότι για τον πολιετή σχεδιασμό και τα τεχνικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το σχέδιο προτάσεων ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σωστές οι προτάσεις της ε, ανακοίνωσής της. Ε, Υπάρχουν άλλα δύο βασικά θέματα. Είναι η πρόσβαση πρώτα απ' όλα στα ύδατα και η κατανομή των αλληλευτικών προσπαθειών. Μιλάμε για τις ημέρες στη θάλασσα, αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε, αλλά όταν εγώ πηγαίνω στην Επιτροπή πει και το συζητώ συνειδητοποιώ ότι σε τοπικό επίπεδο μπορούν, ε, μπορούμε να τα διαχειριστούμε αυτά. Οι κλειστέ ζώνε μπορούν να λειτουργήσουν, οι, οι περιορισμένε ζώνε επίση, ε, η πρόσβαση για τα 12 μίλια, η σταθερότητα, η διαχείριση τη ε, ικανότητα του στόλου. Ναι, εντάξει, αλλά αν δεν ξέρουμε πώ θα τα διαχειριστούμε αυτά σε περιφερειακό επίπεδο, προσοχή, γιατί πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα και αυτό αναφέρεται και σε άλλα σημεία του κανονισμού. Τώρα, ε, τη βάση ε, των διδαγμάτων που αντλήσαμε από τη μεταρρύθμιση του 2002 ε, θα πρέπει να μας απασχολήσει η επιτυχία των Περιφερειακών Ογκομοδοτικών Συμβουλίων. Να ακούσουμε τους ανθρώπους, δηλαδή πέρασαν ένα ηχηρό μήνυμα. Θέλουν τα Περιφερειακά Συμβούλια να έχουν λόγο στην όλη διαδικασία. Θέλουν να επικοινωνήσουν, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σίγουρα λαμβάνεται υπόψη η άποψή τους και με μονόμενα μέλη των ΡΑΚ έχουν πολύ καλέ σχέσει και σε επίπεδο κρατών μελών. Αλλά δεν νομίζω ότι προ το παρόν έχει αναπτυχθεί η σχέση ανάμεσα στα ΡΑΚ και τα ε, πληγόμενα κρατή-μέλη. Διορθώστε με αν κάνω λάθο, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο καλή σχέση. Ε, ποιο είναι το θέμα λοιπόν, ο βασικός στόχος, η συνεργασία, η επικοινωνία, ε, αυτά έχουν τη ζωτική σημασία και να αναρωτιόμαστε με ποιο τρόπο θα λειτουργούσε αυτό στην πράξη. Ακούσαμε πολλά για την ε, νομική πτυχή του ζητήματος ε, και πολλοί τώρα φαντάζομαι μπορούν να υποφεληθούν από μια επανεξέταση αυτών των νομικών επιχειρημάτων, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε μια διευκρίνηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2011 Ευχαριστώ. Ε, είπε ότι η περιφερειοποίηση θα ε, δράζεται στην διακρατική συνεργασία. Αυτή είναι η γενική ιδέα. Ναι, αλλά δεν πρέπει να ε, τυποποιηθεί, να επισημοποιηθεί. Όταν μιλάμε για μακροετή σχεδιασμό, πάλι μιλάμε για τα κράτη-μέλη, αλλά και πάλι εδώ βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα αποφασίσουν, που θα εφαρμόσουν. Οπότε αν μια ομάδα κρατών μελών συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, έχει καλό. Αλλά τι γίνεται στην αντίθετη περίπτωση. Δεν αναφέρεται τίποτα μέσα στο κείμενο. Και αυτό που με τρομάζει ακόμη περισσότερο είναι τι θα σημαίνει αυτό στην ουσία. Δηλαδή, θα έχουμε τη συμφωνία της γαλλιας τη Ιρλανδίας, τη Ισπανία, του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, της ε, Ισπανίας ε, και της Ολλανδίας όπου κάθε κράτος μέλος θα εγκρίνει, περνώντα από το Κοινοβούλιο σταδιακά ένα νέο νομοθέτημα που θα προβλέπει τι θα γίνει σε περίπτωση παρατυπίας ε, τι γίνεται με την ταχύτητα ε, εφαρμογής και μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των γενικών κανονισμών. Δεν θα ισχύουν τα ίδια πράγματα ε, και θα επικρατήσει πλήρες χάος. Είναι σίγουρο αυτό και Μιλάμε για αυτό το θέμα του άρθρου 2. Ε, λοιπόν, εκεί προβλέπεται ότι ε, οι μόνοι που έχουν ε, την αρμοδιότητα είναι τα κράτη-μέλη. Υπάρχει και ο τρίτος δρόμος όμω και ευχαριστώ την νομική υπηρεσία γιατί στη, στο δεύτερο ζήτημα που σχολίασαν να μας έδωσαν μια καλή ιδέα. Ένα λεπτό να περάσω κάποιες διαφάνειες. Έχω υπερβεί ήδη το χρόνο μου, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Λοιπόν, βλέπετε έναν εναλλακτικό τρόπο. Αυτό είναι το σχέδιο της πρότασης ε, που βλέπετε τώρα στην οθόνη. Ε, το κράτος μέλος ε, δύναται να εξουσιοδοτηθεί, να εγκρίνει λέμε. Ε, όπως έχει σήμερα η κατάσταση μπορούμε να προβλέψουμε το εξής σενάριο. Οι τεχνικές λεπτομέρειες μπορούν να αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει πράξη κατεξουσιοδότηση η οποία εξαρτάται από την περιφερειακή δράση των κρατών μελών κατόπιν διαβούλευσης με τα περιφερειακά γνωμοδοτικά ε, συμβούλια. Τι εννοούμε. Ε, είναι σημασιολογική πλέον η συζήτηση. Αφενός έχουμε τα κράτη-μέλη που φοβούνται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θέλουν να αναλάβει με ε, μεγαλύτερη ισχύ από ότι αυτή που προβλέπεται βάσει τη πράξη κατά εξουσιοδότηση. Από την άλλη, στο άρθρο 55.5 παίρνουμε μια έξυπνη απάντηση. Μπορεί να να δοθεί η πράξη κατά εξουσιοδότηση, αλλά υπόκειται σε διάφορα κριτήρια. Και λέμε ότι υπάρχει μια πράξη κατά εξουσιοδότηση, παραμένει ενισχύ εάν το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο δεν αποσύρει την υποστήριξή του για δύο μήνε. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε πράξεις κατά εξουσιοδότηση που να απαιτούν ε, συγκατάθεση από πλευρά αυτών των κρατών μελών που θα έχουν συμφωνήσει για κάποιο θέμα. Δεν πρόκειται για κατάργηση ή για εκχώρηση αρμοδιότητας ε, προς τα κράτη-μέλη τα οποία θα λειτουργούν με χαοτικό τρόπο. Ανταυτού λέμε ότι θα έχουμε ένα περιφερειακό γνωμοδοτικό συμβούλιο που θα επιληφθεί των λεπτομεριών, ε, θα καταλήξουν τα κράτη-μέλη σε συμφωνία, θα την εγκρίνουν και θα υποδείξουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ειδού ε, τώρα μέσω της πράξης κατεξουσιοδότηση θα εφαρμόσετε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατόν αυτό, είναι ε, η προσέγγιση που μας περιέγραψε η, ε, νομική υπηρεσία και έτσι ανακτάται η αξιοπιστία του συστήματος. Αντί να έρχεται ο Ιρλανδός ψαράς και να μου λέει «Μα δεν μπορώ να διαβάσω στα ισπανικά αυτό το σχέδιο, άλλα κάνουν εκείνοι, δεν ισχύουν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού». Ανταυτού λοιπόν θα έχουμε τους ψαράδες κάθε χώρας ε, που θα διαβουλεύονται, θα εκφράζουν άποψή του, θα το λένε στα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη συνέχεια θα θα συμφωνούν ή όχι ε, και στη συνέχεια θα, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει με τις πράξεις κατεξουσιοδότηση την ε, ενωσιακή πλέον νομοθεσία. Αυτή είναι η τρίτη οδός. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κράν. participate in this public hearing. Ευχαριστώ που με επιτρέπετε να συμμετάσχω στην δημόσια ακρόαση και να υποβάλλω τα σχόλιά μου. Ο τίτλος της παρουσίασής μου είναι «Εμπρός στην περιφερειοποίηση» και βασίζεται σε ορισμένες παρατηρήσεις που ακούσαμε και σήμερα το απόγευμα. Όλοι θεωρούμε ότι η περιφερειοποίηση ε, είναι απαραίτητη και όμως δεν υπάρχει σχέδιο δράσης που να οδηγήσει αυτήν. Με την παρουσίασή μου λοιπόν θέλω να συμβάλλω ώστε να παρακινηθούν αυτοί που ασκούν την εξουσία να προχωρήσουν στην περιφερειοποίηση. Θα αναφέρω για ποιο λόγο θεωρώ και πώς μπορεί να γίνει η περιφερειοποίηση και θα έρθω και στην σχέση μεταξύ των οργάνων και της περιφερειοποίησης, δηλαδή των μέσων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και της περιφερειοποίησης. Η κοινή αλληλευτική πολιτική προχωρεί στην τρίτη της μεταρρύθμιση. Όταν άρχισε ο κύκλος των μεταρρυθμίσεων το 2000, της μεταρρυθμίσεων το 2009 ήδη, ήδη οι εφημερίδες έλεγαν ότι οι πολιτικοί λένε ότι έχει αποτύχει η κοινή πολιτική. Σχολιάζω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, είναι ευάλωτη απέναντι σε ε, κριτική όταν λέει ήδη από την αρχή ότι είναι αποτυχία. Γιατί αυτό υπονομεύει την νομιμότητα της πολιτικής αυτής ακόμη περισσότερο. Στη διάρκεια της αξιολόγησης, γιατί αυτό απαιτείται, δεν αρκεί να λένε ότι 88% των αποθεμάτων είναι Πρέπει να δεις ποια πράγματα λειτουργούν και ποια όχι. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να διδαχθείτε και από τις επιτυχίες. Για παράδειγμα, στην Βόρεια Θάλασσα 50 χρόνια ανώτατων ε, επιτρεπόμενων αντιευμάτων και ποσοστώσεων απέδωσαν και επιτυχίες, για παράδειγμα με την ρέγγα και με την χωματίδα. Υπάρχει το πρόβλημα της νομιμότητας. Ως κοινωνιολόγος θα σας πω και πάλι ότι η διαχείριση των ψαριών στην ουσία σημαίνει διαχείριση των εισαγωγικών των ανθρώπων. Πιο σωστό είναι να δώσουμε βάρος στην κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων και επομένως να τους περιλάβουμε στην διακυβέρνηση. Έτσι θα υποφεληθούμε από τις γνώσεις τους, αλλά μπορούμε να τους ζητήσουμε και περισσότερη ανάληψη ευθυνών. Η διαφάνεια αυτή δείχνει την πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Ένα περίπλοκο ε, πεδίο με μια κοινή ε, αλλιευτική πολιτική με διαφορετικέ περιφερειακές θάλασσε, όπου κάθε μια έχει τη δυναμική τη. Χρειάζεται λοιπόν όλα αυτά να ληφθούν υπόψη. Αριστερά βλέπετε την γεωφυσική κλίμακα από τη μια μεριά, από τοπικά οικοσυστήματα μέχρι του ωκεανού και την πολιτικοδιοικητική κλίμακα από την άλλη μεριά, από τι χώρε μέλη μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαίνεται να μην υπάρχει συντονισμό μεταξύ του. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό θέμα αυτό. Εκτός από αυτή την περιπλοκότητα αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο την πρόκληση να περιλάβουμε την αληφτική πολιτική σε ευρύτερες πολιτικές, διότι η πολλαπλή χρήση των θαλασσών μας ε, βάζει ενώπιον νέων προκλήσεων. Και αυτό όμως προσφέρει και ευκαιρίες για να αντιμετωπιστεί το θέμα της περιφερειοποίησης καλύτερα. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε στην διαδικασία της, ε, της θαλάσσιας ότι το να ζητούμε απλώ από τις χώρες μέλη να συνεργαστούν δεν επιτυγχάνει. Άρα, η ε, λύση έγκυται στην περιφερειοποίηση. Τι είναι αυτή η περιφερειοποίηση. Πολλοί ορισμοί ακούστηκαν σήμερα, ωστόσο τρία στοιχεία ακούστηκαν ξανά και ξανά. Πρόκειται για ένα είδος κίνησης. κίνηση προς τα κάτω, αφού άλλωστε η κοινή πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η διαχείρισή της επαφιέται στις χώρες μέλη. Άρα χρειάζεται κίνηση και προς τα πάνω, έτσι ώστε να είναι πιο ε, κομμένες και ραμμένες στις, διάφορες ε, τοπικές συνθήκες η πολιτική. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Μέχρι πού θα πρέπει να φτάσει η κίνηση αυτή. Αυτό θα χρειαζόταν βέβαια πολύ ε, χρόνο να συζητηθεί και έχουν συζητηθεί ορισμένες επιλογές ήδη, αλλά για να συζητηθούν όλα τα μοντέλα και επιλογές, άκουσα βέβαια ορισμένα μοντέλα τα οποία συζητήθηκαν ξανά και ξανά και έχουν αντιμετωπιστεί και στο ερευνητικό πλαίσιο του ΜΕΦΕΠΟ και επίσης στο ΟΝΤΕΜ που ε, αναζητεί μια περιφερειακή προσέγγιση στην αλληλευτική πολιτική. Από αυτά έχουν προκύψει ορισμένε εναλλακτικέ επιλογέ, σε συνεργασία με τις χώρες μέλη αλλά και με τους και με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε από αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Το θέμα του πάνελ είναι για τα όργανα ή τα μέσα που να χρησιμοποιηθούν για την περιφερειοποίηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Η συζήτηση αυτή προέρχεται μάλλον από την μικροδιαχειριστική φύση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, η οποία λέει ότι για να χτυπήσει το καρφί ο ψαράς πρέπει να πάρει το σφυρί. Αλλά γιατί, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τον πέλεκι. Έχει καμία ε, σημασία πώς θα το κάνει. Δικό του θέμα είναι. Τα όργανα ή τα εργαλεία είναι ουδέτερο, έχουν ουδέτερο χαρακτήρα. Μπορεί κανεί να τα πάρει από την εργαλειοθήκη και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλού λειτουργούν καλά, αλλού όχι. Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι η κοινή αλληλευτική πολιτική να κινηθεί προς την κατεύθυνση που οραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δηλαδή μπορεί να στοχεύσει στους στόχους. Και αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία ας δουν πώς, ας αποφασίσουν πώς θα το κάνουν. Τέλος, όπως βλέπετε και στην φωτογραφία αλληγορικά, μπορεί και με τον ένα τρόπο και με τον άλλο τρόπο να καταλήξετε στο ίδιο αποτέλεσμα. Ένα ωραίο σπίτι με μία πισίνα. Πριν να καταλήξω στα συμπεράσματα, θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα από την Βόρεια Θάλασσα, όπου είδαμε τα εξή δύο πράγματα. Πρώτο, η μικροδιαχείριση από πάνω προς τα κάτω, όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν έχει αποδώσει και έχει δώσει ε, κίνητρα στους ψαράδες να ψαρεύουν με μικρότερα μάτια στο δίχτυ και να καταλήγουν επομένως στις απορρίψεις. Ενώ θα έπρεπε να γίνει με διαφορετικό τρόπο και αυτά υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα το Marine Stewardship Council. Το Συμβούλιο παρακολουθεί την βιώσιμη αλία. Ένας, ένα, ε, ο, ολλανδικά σκάφη με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο βγήκαν στη θάλασσα για να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους δίνεται το σήμα του MSC. Χρησιμοποίησαν και το μάτι των 120 συν και το 95 έως 110. Εξήγησαν στο MSC ότι χρησιμοποίησαν το δίχτυ με μικρότερο μάτι μόνο για να μπορέσουν να βγουν περισσότερες μέρες στη θάλασσα. γιατί ο αριθμός των ημερών που τους επέτρεπε το δίχτυο των 120 ήταν πιο περιορισμένος. Πάντως, με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν μικρότερα, μικρότερο ματιού δίχτυα, επομένως τους επέτρεπε αυτό να, ε, να έχουν περισσότερες απορρίψεις. Αυτό είναι που λέγεται το αντίστροφο κίνητρο. Οι ψαράδες είχαν λοιπόν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τα ψάρια αυτά αν μπορούσαν να αποδείξουν δύο πράγματα. Πρώτον, να πείσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποδείξουν ότι την είχαν πείσει ότι ήταν ένα εσφαλμένο κίνητρο το οποίο έπρεπε να αλλάξει και δεύτερον να αποδείξουν ότι τα επίπεδα των απορρίψεων θα ήταν σε βιώσιμο επίπεδο παρόμοιο με αυτό που θα προέκυπτε εάν είχε, είχαν δίχτυα με μεγαλύτερο μάτι. Και μετά από ένα ή δύο χρόνια έπρεπε να γίνει σχετική δοκιμασία. Η MSC έρχεται λοιπόν πάλι στους ψαράδες και ζητάει αποδείξεις. Σε περίπτωση αποτυχίας λοιπόν το σχέδιο διαχείρισης μπορεί να προσαρμοστεί και οι ψαράδες χάνουν το σήμα του MSC εάν δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτές. Αυτό είναι το λεγόμενο result-based management, που είναι αυτό που θεωρούμε ότι χρειάζεται για να γίνει περιφερειοποίηση. Συμπεράσματα. Η διαχείριση των ψαριών στην πραγματικότητα περνάει από την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Βάλτε τους λοιπόν στο παιχνίδι τους ανθρώπους. Θα είναι και καλύτερα τα πράγματα αλλά και πιο νομιμοποιημένα. Επίσης διδαχθείτε και από τις επιτυχίες. Ξεφύγετε από την ιδέα ότι όλα είναι, οδηγούν στην αποτυχία. Υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν σκληρά και έχουν επιτυχίες. Η περιπλοκότητα, η διαφοροποίηση και η δυναμική. Αυτά είναι στοιχεία της αλίας στην Ευρώπη και χρειάζονται λύσεις κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες. πρέπει να μπουν στο μάκρο επίπεδο κάποιες βασικές αρχές και στο μικρό επίπεδο, δηλαδή ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί, ας μείνει σε αυτό το μικρό επίπεδο. Τέλος, η συμμετοχή θα συμβάλλει στην νομοποίηση και στην μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνη. Έτσι λοιπόν, εμπρό προς την περιφερειοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μόνο ο κύριος Γκάλακερ έχει ζητήσει προς το παρόν το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η σημερινή ακρόαση ήταν ε, κάτι που μας επωφέλησε πάρα πολύ. Δεν ε, θέλω να μακρηγορήσω γιατί πρέπει να φύγω. Απλώς ε, ε, ήθελα να αναφερθώ στην μικρή αλία. Έχουμε ένα σκάφος που μπορεί να αρκεί σε μια περιοχή αν είναι εδώ 10 μέτρα, ενώ σε μια άλλη μπορεί να είναι 15. Και σε σχέση με την παρουσίαση που έγινε από τον κύριο Κίτινγκ, Απλώς θα αναφερθώ σε μια περιφέρεια που είναι κοντά στη δική μου χώρα, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την Ορλανδία. Έχουμε το Βέλγιο, την Ολλανδία, τον Μένο Βασίλειο και τη Γαλλία ε, και η δυνάμη του όρθου 17 στην Ιρλανδική θάλασσα, ακόμη και αν έχουμε αυτά τα πέντε κράτη-μέλη που αλλιεύουν, ε, αν υπάρχει περιφερειοποίηση που θα ήταν ευπρόσδεκτη, τελικά θα καταλήξουμε να θέτουμε το ερώτημα, θα έχουμε κάθε κράτος μέλος να εισάγει τη δική του νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν δηλαδή πέντε νομοθετήματα και τι θα γίνει. Θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετική διατύπωση, διαφορετική ερμηνεία και οι ποινέ θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Οι κυρώσεις Θα ήταν αδύνατο λοιπόν αυτό να το ελέγξουμε και να το θέσουμε σε εφαρμογή. Έτσι λοιπόν αντί να έχουμε ίσους κανόνες, ε, έχουμε κάτι που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν αυτό είναι η περιφερειοποίηση, τότε αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν να θέσω το ερώτημα στο κύριο Κίτινγκ. Υπάρχει λύση σε αυτό γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι η Κομισιόν θέλει αυτό. Δεν θέλει πέντε διαφορετικά νομοθετήματα να εισαχθούν σε διαφορετικά κοινοβούλια και σε διαφορετικές κοινωνικέ στιγμέ και θα υπάρχει και πάλι αναθεώρηση θεώρηση της πολιτικής ή θα περάσουν 5-10 χρόνια μέχρι να ε, καταστεί σε εφαρμογή αυτή η νομοθεσία και επίσης ε, το 2002 λέγαμε πολύ συχνά τίποτα δεν συνέβη και τα ΡΑΚ προήλθαν από απόφαση του 2002, λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά, έκαναν κάποιες πάρα πολύ σημαντικές συστάσεις που και το Συμβουλίο και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν δεχτεί τώρα. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό λειτουργήσε όμως. Ε, το αν θα έχουμε περιφερειοποίηση με διαφορετική νομοθεσία και διαφορετική ερμηνεία, αυτό θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή, ίσως είναι κάπως μικροσκελής η ερώτηση, αλλά τέλο πάντων υπάρχει λύση σε αυτό και υπάρχει κάποιο άλλος τρόπος. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στους παρεμβαίνοντες, στους ομιλητές, ε, είτε στην κυρία Κράνη, είτε στον κύριο Κίτη. Και να κλείσουμε. Πρώτα ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ίσως ε, θέλει να επανέλθει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό, αλλά πώς ερμηνεύω εγώ το άρθρο 17 και ολόκληρη την πρόταση έγιος εξή. Ε, τα κράτη-μέλη είναι αυτά που σε εθνικό επίπεδο θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις που απορρέουν από αυτή τη διαδικασία. νομίζω έχει δίκιο ο κύριος Γκάλεχερ. Στην Ιρλανδική θάλασσα θα έχετε πέντε σκάφη δίπλα-δίπλα, το ένα στο άλλο και τελωνιακά θα έχουν την ίδια προσέγγιση, αλλά με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, διαφορετική ερμηνεία των τεχνικών μέτρων κτλ. κτλ. Εγώ αυτό φοβάμαι. Φοβάμαι ε, ότι ε, θα είναι ακόμη πιο άνηση η όρη ανταγωνισμού αντί να επιτύχουμε το αντίστροφο. Αυτό που σας έλεγα με την, τελική, την τελευταία διαφάνεια είναι ότι με μία ε, ίσονο σημασία τροπή τη διατύπωση σε αυτό το άρθρο 17, ε, μία διαχειριστική επιτροπή, ένα διαχειριστικό συμβούλιο, οποιοδήποτε βήμα αυτών των ενδιαφερομένων κρατών μελών ε, θα συνεργάζεται με τα ΡΑΚ και θα καταλήγουν ε, σε, μία, σε ένα κοινό συμπέρασμα, χάρη στο οποίο θα ενεργοποιεί τη διαδικασία της πράξης κατεξουσιοδότησης και θα μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα παραπέμπω και πάλι στο άρθρο 85, όπου ε, προβλέπεται επαρκή προστασία και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο ε, για να εξασφαλίσουν ε, την ορθή λειτουργία τη διαδικασία. Δηλαδή, με αυτή την αλλαγή τη διατύπωση θα έχετε την επιλογή του σωστού επίπεδου λήψη απόφαση πέρα από την εφαρμογή. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κρά. Θέλετε το λόγο. Thanks. Όχι, όχι, ευχαριστώ, λέει η κυρία Κρά. Εσεί και τη Επιτροπή. Ο Πένα, σε ευχαριστώ. Θα κάνω δύο διευκρινήσει. Καταρχήν, πράγματι ότι πρέπει να καταστεί πολύ το σαφέ ότι για την Κομισιόν είναι σημαντικό και πρέπει η Κομισιόν να κάνει οποιαδήποτε πρόταση να ε, λάβουμε υπόψη την άποψη τόσο του ISIS, τόσο και του ΣΤΕΦ, δηλαδή της επιστημονικής κοινότητας, αλλά επίσης θα πρέπει να, να συμβουλευτούμε και τα ΡΑΚ. Ε, η υποχρεωτική διαβούλευση με τα αρμόδια ε, επιστημονικά όργανα και με τα ΡΑΚ δεν ε, αναφέρεται κάπου, αλλά η Κομισιόν ε, θέλει να το κάνει. Εγώ νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει καμία απόκληση επί της ουσίας. Όλοι θέλουμε οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν ε, να γίνονται με μια προηγούμενη διαβούλευση των επιστημονικών οργανών και των ΡΑΚ. Είναι απόλυτα σαφές αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε μια λύση που από νομική σκοπιά να ικανοποιεί ε, και τις νομικές υπηρεσίες των θεσμών. Δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα βέβαια για το θέμα αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. κατόπιν σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κίντιν και ο κύριος Γκάλακερ η ιδέα είναι ότι πράγματι το μοντέλο που προτείναμε είναι ένα μοντέλο το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να υιοθετούν εθνικέ νομοθεσίε για να μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή τι μεγάλες αρχές που έχουν υιοθετηθεί από το συνομοθέτη. Και γνωρίζουμε ότι εδώ έχουμε τον κίνδυνο, τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν αυτές τις εθνικές νομοθεσίες ε, με έναν τρόπο όχι ακριβώς ισόδυναμο ή σε διαφορετική χρονική στιγμή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή υπάρχει κίνδυνος αυτός, προβλέψαμε ένα μηχανισμό νομικό και κατόπιν έχουμε και ένα μη νομικό μηχανισμό, ένα πολιτικό μηχανισμό διαπραγμάτευση. Το επιχείρημα το νομικό είναι ότι έχουμε προβλέψει δυνατότητα, αν τα κράτη-μέλη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για το με το ποιο τρόπο θετήσουν τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί μέσω τη εθνική νομοθεσία, ε, πάντοτε μπορεί να παρέμβει η Κομισιόν. Η Κομισιόν εκεί θα είναι πάντα για να επιλύσει το πρόβλημα, αν τα κράτη-μέλη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν ή αν δεν ε, μπορέσουν να υιοθετήσουν εθνικά μέτρα γέρος. Αυτός ο μηχανισμός έχει προβλεφθεί. Και θέλω να σας ανακοινώσω ότι η ιδέα ότι η Κομισιόν μπορεί να, το, να μπορεί να το κάνει αυτό δεν γίνεται και πολύ ε, θετικά αποδεκτή από το Συμβούλιο. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι απόπειρα της Κομισιόν να κερδίσει ε, αρμοδιότητες, να ενισχύσει την εξουσία της, αλλά δεν ισχύει. Και ο άλλος μηχανισμός, ο πιο πολιτικός είναι ότι φυσικά Πρέπει να υπενθυμίσω ότι ε, θα λάμβανε χώρα η λήψη της περιφερειμένης απόφασης όταν το συναποφασίσουν οι συνομοθέτες ανά περίπτωση. Και φυσικά, όταν οι συνομοθέτες αποφασίσουν ότι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση κάποια μέτρα θα μπορούσαν να θετηθούν από τα κράτη-μέλη, θα το έκαναν με... γνωρίζοντας ε, το βαθμό της πολιτικής βούλησης ε, αυτών των κρατών μελών για να συμφωνήσουν. Έτσι λοιπόν εσείς οι ίδιοι συνομοθέτες θα συμφωνούσατε στο να δώσετε αυτή την αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν ορισμένα ζητήματα μόνο στις περιπτώσεις που εσεί οι ίδιοι θα βλέπατε αν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση συμφωνίας ή όχι και αυτή η ικανότητα για να γίνει συντονισμένα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο, η κυρία Ρόντου για να κλείσετε. Ναι, ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το σημερινό απόγευμα. Νομίζω ότι διδαχθήκαμε πολλά από τις απόψεις των διαφόρων ε, συνομιλητών μας και νομίζω μάλιστα ότι έτσι ήρθησαν και ορισμένα εμπόδια. Όλοι νομίζω εδώ συμφωνούμε ότι θέλουμε μια καλύτερη αλληλευτική πολιτική, περισσότερο υπεύθυνη. Νομίζω μάλιστα ότι η ε, υφιστάμενη αλληλευτική πολιτική από πολλούς κρίθηκε ως αποτυχία. Η γνώμη μου είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουμε διαφορετικούς κανόνες για την αλία, αλλά να επιτύχουμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο που να είναι τόσο στέρεο, ώστε από τη μια μεριά να μην υποσκάπτεται η ισχύση του ευρωπαϊκού δικαίου, από την άλλη μεριά να υπάρχει και η απαραίτητη περιφερειοποίηση. Έτσι ακούστηκαν σήμερα πολύ καλές ιδέες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, να περιληφθούν ενδεχομένως στον βασικό κανονισμό ή στην περαιτέρω παράγωγη νομοθεσία αργότερα. Να εξετάσουμε μαζί με ποιον τρόπο θα οργανώσουμε καλύτερα τα πράγματα. Θα μελετήσω πολύ προσεκτικά τα έγγραφα που υποβάλλατε και αν έχετε και άλλες ιδέες είμαι ανοιχτή. Πολύ ευχαρίστως να τις δεχθώ, να μου τις αποστείλετε και αφού σας ευχαριστήσω και πάλι, εκφράζω την ελπίδα ότι όλοι θα επιστρέψουμε στην βάση μας με το αίσθημα ότι όντως έχουμε κάνει ένα βήμα προς περισσότερη συνεργασία υπέρ της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ε, τι τις ευχαριστίες κυρίως προς τους και βεβαίως και προς όλους τους βουλευτές που έλαβαν το λόγο ξεκαθαρίστηκαν πολλά θέματα. Σήμερα παραμένουν βέβαια και άλλα που πρέπει να ξεκαθαριστούν. Έχουμε ακόμα πολλή συζήτηση μπροστά μας, διότι το μέρος αυτό της συζήτησης, της μεταρρύθμισης μάλλον, θα πρέπει να υλοποιηθεί. Θα διαρκέσει η συζήτηση αυτή ακόμα πολλές εβδομάδες και μήνες και οι ακροάσεις αυτές που γίνονται με εμπειρογνώμονες όπως εσείς είναι πάρα πολύ σημαντικές. Με στόχο να υπάρξει το καλύτερο, το βέλτιστο δυνατό έγγραφο στο τέλος της προσπάθειας αυτής. Ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε τον πρόεδρο. Αύριο συνεχίζουμε στις 9 το πρωί.